Is it working now? It's okay. Yeah. It's okay. Va bene. Allora, λοιπόν. riprendiamo i lavori adesso. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Ε, λύθηκε το τεχνικό πρόβλημα. Νομίζω ότι ακούγεται η διερμηνία. Λοιπόν, πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη, έγκριση του σχέδιου ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θεωρώ ότι εγκρίθηκε. Σα παρακαλώ, συνάδελφοι. Ε, Szanowna Pani Przewodnicząca, e, ja zwrócić uwagę na... Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι για μια συγκεκριμένη αναφορά 192 του 2009 και το σημείο 65 της ημερήσιας διάταξης που είναι στον κατάλογο των σημείων Β προτείνω να μην την κλείσουμε αυτή την αναφορά Πιστεύω ότι δεν είναι επαρκή η διευκρινή τη Επιτροπή και θέλω να συνεχίσουμε τη συζήτησή μα για την αναφορά αυτή. Ναι, ναι, ε, Πολύ ωραία. Μα άλλωστε ήδη είχα ενημερωθεί για το θέμα αυτό. Στο παράδειγμα Β, εκεί που έχουμε τις ε, προτάσεις ε, για τις ε, προτάσεις που διπώθηκαν στη Γενική Γραμματεία, προσθέτω ότι υπάρχει και μια άλλη επισήμανση για τη 0439 του 2009 και για τις δύο έχουμε αίτηση να, κρατήσουμε, να τις κρατήσουμε ανοιχτές. Άρα να εξακολουθήσουμε να τις ε, εξετάζουμε. Λοιπόν, κατά τα άλλα, δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Υπάρχει πρόβλημα. Συγγνώμη. Δεν, δεν, καταλάβα, δεν κατάλαβα, το λόγο. Σε το συγγνώμη, ωραία. Λοιπόν, θεωρούμε ότι ανακρίθη η μερίσια διάταξη, η ημερήσια διάταξη. Δεύτερο θέμα, έγκριση των πρακτικών Τη συνεδρίες τη 1 Οκτωβρίου και τη 19 Οκτωβρίου. Και ε, έχουμε και τον κατάλογο των ε, παραδεκτών αναφορών που έχει, έχουν προσαρτηθεί στα ε, δύο αυτά πρακτικά. Αν δεν έχετε αντιρρήσει, θεωρούμε ότι και τα πρακτικά και τα παραρτήματα εγκρίθηκαν από την Επιτροπή μας. Τρίτο θέμα. Θα ήθελα να σας πω ότι όσον αφορά τη Σύνοδο του Δεκεμβρίου θα έχουμε τους αναφέροντες, ε, όχι, ε, την, τη συνεδρίαση, τους ε, αναφέροντες στο 9, 10, 11, 12 και 15. Σα προσθέτω ω ανακοίνωση ότι το έγγραφο που αφορά τις αναφορές που θα κλείσουν ή που θα επανανοίξουν, ε, το πήρατε. Δεν, έχω, δεν έχουμε λάβει καμία παρατήρηση. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι κρίση Με τη μορφή αυτή που το πήρατε. Αν δεν έχετε αντιρρήσει και όσον αφορά το σημείο αυτό, θεωρώ ότι εγκρίθηκε η πρόταση. Επίσης να σας πω και σίγουρα θα διαβάσατε τον κατάλογο των νέων των υποψήφιων νέων επιτρόπων. Ιδιαίτερα όσον αφορά το σημείο αυτό, να σας πω ότι εμείς εδώ και καιρό προετοιμαζόμαστε για την, να ζητήσουμε ε, ακρόαση επιτρόπου ε, αρμόδιο για τα δικά μας θέματα, ε, πράγμα σχετικά καινούριο. Και από ό,τι φαίνεται θα γίνει η ακρόαση αυτή με τον Επίτροπο Μάρο Σεφκόβιτς, που είναι ο Επίτροπος Αντιπρόεδρος, ε, που είναι υπεύθυνο για θεσμικά ζητήματα και, θέματα, και διοικητικά. Αλλά εδώ ήθελα να σε επιστήσω την προσοχή στο εξής. Η κυρία Βιβιάν Ρέντιν και αυτή η αντιπρόεδρος είχε ως αρμοδιότητα τα θέματα δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ηθαγένειας. Όσον αφορά το σημείο αυτό, σας υπενθυμίζω, αν τυχόν το δυσμονήσατε, ότι κατά την ε, συνεδρία της επανεκλογής του κυρίου Μπαρόζο, ε, ζητήσαμε εξ ονόματος της Επιτροπής από τον ε, πρόεδρο Μπαρόζο να προσέξει ιδιαίτερα ε, τις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας και να υπάρξει ε, επίτροπος, υπεύθυνος. Τότε, απαντώντας στην παρέμβασή μου, ο κύριος Μπαρόζος μου είπε ότι όσον αφορά τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών, θα ανέθετε στον αρμόδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, για τη δικαιοσύνη και την ηθαγένεια επίτροπο και τα θέματα της δικής μας Επιτροπής. Το είχε, μου είπε, ήδη σκεφτεί και επιβεβαίωσε τις προθέσεις του όταν εγώ του έκανα τη σχετική ερώτηση. Ήθελα λοιπόν να σας θέσω αυτό το θέμα και νομίζω ότι εμείς ως Επιτροπή πρέπει να ζητήσουμε την ακρόαση ε, της Επιτρόπου Ρέντιν. Από ό,τι φαίνεται όμως και βλέποντας και το έγγραφο της ε, Διεύθυνσης του Κοινοβουλίου βλέπω ότι εδώ αναφέρεται ο Επίτροπος Ευκόβιτς. Αν συμφωνείτε θα ε, επαναλάβω για άλλη μια φορά το αίτημα για συμμετοχή στην ακρόαση της κυρίας Ρέντιν. Θέλετε το λόγο, κύριος Μπουσούτη. Yes, thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι πρέπει οπωσδήποτε να συμμετάσχουμε στη διαδικασία ακρόασης ε, της Επιτρόπου Ρέντινγκ που θα είναι και αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Από ό,τι γνωρίζω, οι αρμοδιότητες της θα συμπεριλαμβάνουν και την ηθαγένεια και την ε, επικοινωνία. Άρα νομίζω ότι ακριβώς η κυρία Ρέντινγκ είναι η επίτροπος με την οποία πρέπει να κάνουμε ακρόαση. Θα πρέπει και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ βέβαια να συμμετάσχει στην ακρόαση για την Επίτροπο, αλλά νομίζω ότι η Επιτροπή Αναφορών πρέπει να συμμετάσχει σε αυτή την ακρόαση της ε, κυρίας Βιβιάν Ρέντινγκ. Είναι ακριβώς ο τομέας ενδιαφερόντων της Επιτροπής μας. Και να σας πω την αλήθεια, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να έχουμε ακρόαση και με τον άλλο επίτροπο που είναι υπεύθυνο θεσμικών θεμάτων. Εμείς ως Επιτροπή Αναφορών περισσότερο ενδιαφερόμαστε για τα θέματα των πολιτών και των ε, ανακοινώσεων της Επιτροπής. Γιατί λοιπόν έχουμε ακρόαση με τον κύριο Σεύκοβιτς. Ίσως ο λόγο είναι ότι δεν υπήρχε άλλη επιτροπή και κάποια επιτροπή έπρεπε να κάνει ακρόαση με τον κύριο Σεύκοβιτ. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι επαρκή λόγο. Εγώ είμαι λοιπόν, λοιπόν κυρία Πρόεδρε, υπέρ τη θέση ότι θα πρέπει η επιτροπή μα να συμμετάσχει στην ακρόαση τη κυρία Βιβιάν Ρέντινγκ και ακριβώ όπω σα είπα γιατί καλύπτει τα θέματα ηθαγένεια και επικοινωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Όκεν. Κυρία Όκεν. Ευχαριστώ. Συμφωνώ, Πρόεδρε, με αυτά που είπατε μου έκανε εντύπωση, δεν φορούσατε τα ακουστικά σα και νόμιζα ότι καταλαβαίνετε τα δανέζικα. Λοιπόν, τώρα που φοράτε και τα ακουστικά σας, να σας ξαναπώ ότι συμφωνώ σχετικά με την συμμετοχή της Επιτροπής μας, ε, γιατί και εγώ έχω προσπαθήσει πάρα πολύ ε, να κάνουμε την Επιτροπή μας μια Επιτροπή που θα είναι γνωστή ως Επιτροπή που έχει σχέση με τον πολίτη και τα θέματα των πολιτών. Νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να δούμε και τον Επίτροπο Αρμόδιο για το Περιβάλλον, γιατί αν δούμε πόσο χρόνο δίνουμε για περιβαλλοντικά θέματα, νομίζω ότι και με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος θα πρέπει να κάνουμε ακρόαση. Και όταν κάναμε την έκθεσή μας για το Natura 2000 και εξετάσαμε τα θέματα της οδηγίας, ε, μας απασχόλησε πάρα πολύ το περιβάλλον. Βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε με όλους τους επιτρόπους ακρόαση, αν έχουμε μόνο δυνατότητα για έναν επίτροπο, θα πρέπει την επίτροπο που είναι υπεύθυνη για θέματα πολιτών να δούμε. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Κυρία Βόλης. Απλά θα ήθελα και εγώ να προσθέσω τη φωνή μου σε εκείνους που υποστηρίζουν ότι αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να έχει κάποια κρόση με την κυρία Ρέντινγκ. Παρά το γεγονός ότι νομίζω το πρόβλημα θα είναι το εξής. Η κυρία Ρέντινγκ έχει ένα τεράστιο χαρτοφυλάκι, όχι μόνο καλύπτει ε, τους πολίτες και την επικοινωνία, αλλά καλύπτει όλο τον κλάδο της ε, αστικής δικαιοσύνης, ε, που είναι ο τομέας της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και καλύπτει τα δικαιώματα που είναι της Επιτροπής Live. Συνεπώς αυτή η κυρία έχει πολλά να κάνει και φαντάζομαι ότι όταν είχε σκεφτεί το Κοινοβούλιο να χωρίσει τα χορτοφυλάκια δικαιοσύνη, δεν είχε σκεφτεί ότι θα χωριστεί με αυτόν τον τρόπο. Διότι τελικά ε, ένα άτομο, μία επίτροπο έχει πολύ ε, βάρος. Βεβαίως, νομίζω ότι αυτό που είπε ο κύριος από τη Σλοβακία, δεν ξέρω πολύ καλά πώς να προφέρω το όνομά του, νομίζω ότι έχει δίκιο, αλλά θα έχει εκείνο νομίζω ε, την αρμοδιότητα για τη διαφάνεια, συνεπώς για τον ε, Ευρωπαίο Συνήγορο και οτιδήποτε έχει σχέση με τα όσα κάνουμε εδώ. Ευχαριστώ. Sí. Επίτροπος για, δικαιοσύνη, για, τις δικαιοσύνη, για τη δικαιοσύνη της ελευθερίας των πολιτών και την, ε, ε και την Ιθαγένεια είναι επιτροπές σε Λίμπε, Γιούρι, Φαμ και Κάλτσουρ για όλες αυτές τις επιτροπές. Από την άλλη, όσον αφορά το φόρτο εργασίας του συγκεκριμένου επιτρόπου, αν επιτρέπετε να σταθώ για λίγο, ο Επίτροπος υπεύθυνος για τα θεσμικά θέματα Ε, συνδέεται με την ε, ε, ΑΦΚΟ, Γιούρι, Budget και Πέτη. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν νομίζω, μία ή άλλη είναι τα δύο πράγματα. Για λόγους λοιπόν που έχουν να κάνουν την ουσία. Δηλαδή εγκύτητα με την ουσία των θεμάτων που μας απασχολούν και με τα δικά μας καθήκοντα. Εμείς θα μπορούσαμε λοιπόν, χωρίς να διαταράξουμε ιδιαίτερα το φόρτο εργασίας των επιμέρους επιτρόπων, θα μπορούσαμε να επιμείνουμε σε αυτό το αίτημα το οποίο νομίζω ότι, ε, με το οποίο νομίζω ότι συμφωνούν οι περισσότεροι συνάδελφοι. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπε η κυρία Όκεν, τώρα, να φανταστούμε ακροάσεις ε, τον, ε, με τον ε, Επίτροπο για το Περιβάλλον, ε, ε κοιτάξτε, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να, έχουμε, να συνδεθούμε με τις ακροάσεις όλων των Επιτρόπων. Κοιτάξτε, λόγω των ε, αρμοδιοτήτων μας, εμείς εκ των πραγμάτων ασχολούμαστε με, με όλα τα θέματα. Με, και σίγουρα θα πρέπει τότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μιλήσουμε και για να, να συμμετάσχουμε και στην ακρόαση Επίτροπο Εσωτερική Αγορά, μεταφορέ πάρα πολλά θέματα που αφορούν τις μεταφορές που μας απασχολούν. Άρα, να εστιάσουμε την προσοχή μας. Τουλάχιστον να κερδίσουμε ένα εκπρόσωπό μας, αν θέλετε, δόση τη Επιτροπής και μετά με τους υπόλοιπους θα έχουμε σχέσεις ε, ε, ανάλογα με τα θέματα τα οποία θα μας απασχολούν σε επιμέρους αναφορές. Ντεμπρούν. Συνάδελφος κυρία Ντεμπρούν. Ευχαριστώ. Θα επαναλάβω, δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα υπόθηκαν, απλά θα ήθελα και εγώ να υποστηρίξω ε, τις προτάσεις που κάνατε σχετικά με την ακρόαση τουλάχιστον σε ό,τι έχει σχέση με την ακρόαση κύριε Ρέν. Εντάξει. Απλά και εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω την πρότασή σας. Αυτό ήθελα να πω, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ. Συγγνώμη, ε, μου διέφυγε ένα λεπτό η προσοχή. Ε, ο Ντέβιντ Λό μου υπεδείκνυε να σας υπενθυμίσω αυτό το θέμα με τις ερωτήσεις που είχαμε διατυπώσει για τις ακροάσεις. Ε, επειδή τώρα πλησιάζει η ημερομηνία, ο Γενάρης φτάνει όπου θα γίνουν αυτές οι ακροάσεις. Σας καλώ λοιπόν να ξαναδούμε ενδεχομένως αυτές τις ερωτήσεις. Για να δούμε, είναι εντάξει, μήπως πρέπει να συμπεριλάβουμε και νέα θέματα, τα οποία τυχόν σε απασχολούν. Όσον αφορά λοιπόν το σημείο αυτό, νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο και πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσια διάταξης. Και prevede già la prima petizione, entriamo nel settore ambiente, apriamo... Λοιπόν, πάμε στον τομέα περιβάλλον, ε, στο τμήμα Α της ημερήσιας διάταξης, 251 του 2007, Μαρίν Γκαλέα, της Μαρίν Γκαλέα. Η αναφέρουσα δεν είναι παρόν. Εκ μέρους της Επιτροπής, η Φρανσουάς Κρέμερ είναι υπεύθυνη. Έχετε το λόγο. thank you, Mrs. Ο κύριος, συγγνώμη. Δεν είμαι η Φρανσουάζ Κρέμερ, και δεύτερος στον κατάλογο. Θα καλύψω και τα δύο θέματα, τις δύο αναφορές που αφορούν ε, το ίδιο σημείο στη Μάλτα, στη Μάλτα στην Ίσο Γκόζο, το, την περιοχή Τατζέν. Η δεύτερη αναφορά είναι η παριθμόν 10-10 και έχει σχέση με το αν αυτή η περιοχή εντάσσεται στο Natura 2000 και το δεύτερο θέμα που καλύπτει η πρώτη αναφορά έχει σχέση με πιθανή ζημία που επιφέρει σε αυτό το χώρο η ανάπτυξη ενός τουριστικού προγράμματος για την περιοχή. Όσον αφορά το αν θα συμπεριληφθεί η Επιτροπή στο δίκτυο Natura 2000, πρέπει να πω ότι οι αρχές της Μάλτας έχουν θέσει αυτή την περιοχή στην οδηγία για τους οικοτόπους και υπάρχει και άλλο ένα ζήτημα, ορισμός αυτής της περιοχής ως, περιοχή, ως ζώνη ειδικής προστασίας σύμφωνα με την οδηγία των πτηνών. Η Επιτροπή είχε αρχίσει μια διαδικασία παραβάση κατά της Μάλτας πριν από χρόνια για ανεπαρκή ορισμό ζωνών ειδικής προστασίας για την προστασία των πτηνών τη. και μετά τον ε, ορισμό αυτής της περιοχής ως ιδιάζουσα σημασίας, αυτή η υπόθεση παράβασης έκλεισε πλέον Στι αρχέ του 2009 την έκλεισε αυτή την υπόθεση η Επιτροπή. Όσον αφορά το ΤΑΣΕΝΚ, αυτό το συγκεκριμένο χώρο που αναφέρεται, τμήμα αυτού του χώρου ήδη έχει οριστεί ω ζώνη ειδική προστασία, όμω ε, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα που έχουν υποβάλει οι αρχές της Μάλτας, και βάσει της ανταλλαγής πληροφοριών που είχαμε με τις αρχές της Μάλτας, φαίνεται ότι ο, ο χαρακτηρισμός αυτής ε, της ε, περιοχής ε, έχει ανεπαρκή δεδομένα σύμφωνα με την οδηγία για τα πτηνά και τα στοιχεία τα οποία δίδονται για τους κρυμνούς στις παράκτιες περιοχές επίσης δεν είναι επαρκή. Ίσως ε, οι αναφέροντες ανησυχούν περισσότερο για το δεύτερο θέμα που αφορά την οδηγία των πτηνών και την ε, προτινόμενη επέκταση ενός ε, ξενοδοχείου και, την, και ένα πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης για την περιοχή. Η Επιτροπή έχει συζητήσει το θέμα αυτό με τις αρχές της Μάλτας αρκετές φορές και όπως είχαμε πει και σε μια προηγούμενη παρουσίασή μας στην Επιτροπή σας, Θίξαμε και πάλι το θέμα στην ετήσια συνάντηση με τις αρχές της Μάλτας σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δοθεί, φαίνεται καταρχήν ότι η αρχική αίτηση Γι' αυτό το πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης απερίφθη από τις αρμόδιες αρχές που έδωσαν αρνητική γνωμοδότηση για την ε, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είχαν γίνει για αυτό το πρόγραμμα. Παράλληλα υπάρχει και κάποια νομική διαδικασία που έχει ξεκινήσει στη Μάλτα κατά του προγράμματος αυτού. Στη συνέχεια οι αρχές της Μάλτας <coughs> ζήτησαν ε, ένα νέο σχεδιασμό αυτού του προγράμματος ε, για να μην ε, είναι επιζήμιο προς τις περιοχές Natura 2000 του Τασέγκ και φαίνεται ότι ήδη έχει σχεδιαστεί αυτό το πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης διαφορετικά πλέον θα γίνει μια επικαιροποιημένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η αξιολόγηση με βάση το άρθρο 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους θα γίνει εκ νέου πριν ληφθεί τελική απόφαση. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλουμε να υπάρχει πλήρης επιστημονική αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων επί αυτού του χώρου, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο το πρόγραμμα ανάπτυξης, αλλά ε, και όλα τα άλλα, όλες τις άλλες παραμέτρους σωρευτικά. Και δεύτερον, ζητήσαμε γραπτός να γίνει μια επικαιροποίηση της εξέτασης από τις αρχές της Μάλτας σχετικά με τη λήψη αποφάσεων για αυτό το πρόγραμμα. Και αυτό σημαίνει ότι όταν θα έχουμε τις επικαιροποιημένε περιβαλλοντικές επιπτώσεις, θα προωθηθούν από τις αρχές της μάλτα στην Επιτροπή και η Επιτροπή από αυτής της θα αναλύσει την κατάσταση για να αξιολογήσει αν υπάρχει παραβίαση κοινωτικής νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Uh, yes, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σα ευχαριστήσω που περιλάβατε αυτό το σημείο στην ημέρα διάταξη τόσο γρήγορα μετά από την τελευταία συνεδρίαση που είχαμε. Επίση, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τι πληροφορίε που μα έδωσε. Θα ήθελα μια διευκρίνηση από την Επιτροπή, αν κατάλαβα καλά την θέση τη. Αν κατάλαβα λοιπόν καλά, δεν υπάρχει παραβίαση με βάση ε, την κατάσταση της περιοχής, ε, δηλαδή ε, το καθεστώς της, πώς έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα με τον, την κοινωτική νομοθεσία. Δεύτερον, δεν είναι ακόμα σαφές κατά πόσον υπάρχει παραβίαση όσον αφορά το προγραμματιζόμενο τουριστικό πρόγραμμα, το project. Κατάλαβα καλά. Πρώτα να μου πείτε, να μου δώσετε αυτή τη διευκρίνηση και μετά θα συνεχίσω. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που να θέλουν το λόγο, διαφορετικά να δώσω... Ε, α, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ναι, σωστά καταλάβατε. Δεν υπάρχει παράβαση σχετικά με το χαρακτηρισμό της περιοχής και με το βιότοπο, δηλαδή την οδηγία ε, για τον ε, βιότοπο για τα πουλιά. Και δεύτερον, όπως σας είπα, ναι, έχει κλείσει επειδή υπήρχαν ορισμένα ευαίσθητα είδη και όσον αφορά τώρα ε, τη συγκεκριμένη τουριστική ανάπτυξη. Και εδώ δεν υπάρχει καμία παραβίαση κανόνων επειδή δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία απόφαση. Και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο στάδιο της αξιολόγησης για να δούμε κατά πόσον οι μελέτες ε, περιβαλλοντικού αντικτύπου θα επικαιροποιηθούν και κατά πόσον αρκούν ή όχι. Τη στιγμή που θα έχει δει αυτές τις μελέτες ε, η Επιτροπή, τότε θα αποφασίσει τι συνέχεια θα δοθεί σε αυτή την υπόθεση. ό,τι. Λοιπόν, με βάση την απάντηση που μου δόθηκε, αυτό που με απασχολεί, κυρία Πρόεδρε, είναι το εξή. Αυτό το θέμα θα έπρεπε να κλείσει το ταχύτερο δυνατόν. Δεν θα ήθελα να προδικάσω το αποτέλεσμα, διότι θα εξαρτηθεί από την απάντηση που θα δώσουν οι αρχές της Μάλτας. Αν κατάλαβα καλά, οι αρχέ τη Μάλτας μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου έχουν δώσει ως προθεσμία για να δοθεί η απάντηση και κατόπιν η Επιτροπή θα μπορέσει να δει κατά πόσον υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας ή όχι. Αυτό που ασχολεί έχει περισσότερο σχέση με το χρόνο. Αυτή είναι μια αναφορά που έχουν υπογράψει 10.000 άτομα και για μια χώρα του μεγέθους ηθικής μου ο αριθμός αυτός είναι σημαντικό. Πιστεύω λοιπόν ότι η υποβολή αυτή τη αναφορά ε, το 2007, το γεγονό ότι υπευλήθη το 2007, πριν από δύο χρόνια, ε, πιστεύω ότι πρέπει να τους δοθεί μία σαφής απάντηση, ναι ή όχι. Κατά πόσον η σημερινή κατάσταση ως έχει συμφωνεί με την κοινοτική νομοθεσία ή όχι. Αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε ε, στους ανθρώπους που υπέγραψαν Εν κατακλείδη, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σα παρακαλέσω να παραμείνει αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη, διότι χάρη στο γεγονό ότι παραμένει στην ημερήσια διάταξη, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προωθούν αυτό το θέμα για να καταλήξει προ την άκρη τη δίτα κατεύθυνση. Συνεπώ, διατηρώντα την ημερήσια διάταξη αυτό το θέμα, στην ημερήσια διάταξη βοηθάμε του πολίτε που, που έχουν καταθέσει αναφορά να πάρουν μια απάντηση. Πολύ καλά, σα κατάλαβα. Κατάλαβα τι θέλετε. Δηλαδή να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά, ώστε με αυτόν τον τρόπο να επιταχύνουμε τη διαδικασία, κυρίως σε ό,τι αφορά την απάντηση που αναμένει η Επιτροπή από τις Μαλτέζικες Αρχές. Για τα τουριστικά projects. Συνεπώς πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά όπως και η Επιτροπή, αναμένουμε τις απαντήσεις των αρχών της Μάλτας και τότε θα δούμε τι μέτρα θα πάρουμε στην Επιτροπή μας. Λοιπόν, αυτές οι δύο αναφορές θα παραμείνουν ανοιχτές. Ξέχασα τη δεύτερη όμως. Μας είπε η Επιτροπή ότι ε, και αυτή καλύπτονταν. Ερχόμαστε στην αναφορα 87, 687-2008 που υπέβαλε ένας ε, πολίτης μαλτέζικης ηθαγένειας. Ο αναφέρον δεν είναι παρόν. Παρακαλώ, το λόγο Επιτροπή. Sorry, you have missed. Ζητώ συγγνώμη, ο κύριος Φέγγσταρεν από την Επιτροπή είναι εδώ. Ίσως θα έπρεπε να ξεκινήσω με τη δεύτερη, διότι όλο το πρόβλημα με τη μεταφορά αυτής της οδηγίας στη Μάλτα ξεκίνησε με το γεγονός υπήρχαν καταγγελίες από ε, την ε, αρχές η 275-2006 όσον αφορά τη δικασία παραβίαση το 2008 οι Μαλτέζικες αρχές τροποποίησαν τη δημοθεσία τους και άρχισαν να ρυθμίζουν την ε, κατάσταση ε, των γραμματέων διεύθυνσης των τοπικών συμβουλίων. Η πρώτη ε, αναφορά δεν αναφέρει τους γραμματεί διεύθυνση, αλλά ενός δασκάλου, ο οποίος αισθάνεται ότι υπήρχε διακριτική μεταχείριση εναντίον του, διότι αντιθέτω προς τους γραμματεί τη διεύθυνση, η σύμβασή του δεν μετατράπει σε ε, απεριορίστου χρόνου σύμβαση. Αλλά άλλαξε η νομοθεσία της Μάλτας και κατά πόσον υπάρχει ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με ε, την οδηγία είναι ένα θέμα το οποίο θα αποφασίσουν τα εθνικά δικαστήρια. Και αν ο αναφέρον θεωρεί ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση εναντίον του, τότε θα έπρεπε να στραφεί στα εθνικά δικαστήρια. Όσον αφορά αυτή την υπόθεση σε κρεμότητα, υπογραμμίζω ότι παρά το γεγονό ότι είναι ανοιχτή υπόθεση, δεν συνδέεται με του υπενιγμούς που έκανε ο αρχικό αναφέρον όσον αφορά ε, ότι είναι ένα ξεχωριστό θέμα. Είναι ξεχωριστό θέμα και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω. Απαντήσατε και για τις δύο αναφορές ή για τη μία για τις δύο. Δεν κατάλαβα. Το κύριο Άντριαν Μιφσούντ, 275-2006. Γι' αυτό απαντήσατε. Ξεκίνησα με τη 275 και καταλήγω στο 27-2008 διότι ξεκινάμε με την αλλαγή της νομοθεσίας που έχει σχέση με τη δεύτερη αναφορά. Number seven. Η επτά ήταν η αναφορά που βρισκόταν ε, στην αρχή της διαδικασίας παραβίασης, αλλά μεταξύ άλλαξε νομοθεσία. Και η 87 ε, αντίθετα με τους γραμματείς διεύθυνση των τοπικών συμβουλίων, ε, αφορά έναν δάσκαλο και νομίζω ότι ε, θεωρεί ότι έπρεπε η νομοθεσία να είχε εφαρμοστεί για αυτόν και δεν είχε γίνει. Και αυτό το θέμα συνεπώ έχει παραμείνει ανοιχτό. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε αν δημιούργησα παρεξήγηση. c'è anche una parte di responsabilità nostra, quindi le due petizioni sono collegate. Λοιπόν, συνδέονται μεταξύ τους αυτές οι δύο αναφορές, εντάξει. Ξεκινάμε λοιπόν από ε, την ε, αναφορά του σημείου 7. Θα τις δούμε μαζί, είπατε. Ευχαριστώ. Συμφωνώ, είναι αλληλένδετες οι δύο αναφορές, ναι. Αφορούν την ίδια οδηγία, γι' αυτό. Συνεπώς είναι αλληλένδετες αλλά δεν με έχει ικανοποιήσει η απάντηση της Επιτροπής παρόλα αυτά. Γιατί? Η 12.87.2008 η 87 Η σχέση με το κατά πόσον έχει μεταφερθεί την εθνική νομοθεσία σωστά η οδηγία αν κατάλαβα καλά, μια διαδικασία παραβίασης παραμένει σε κρεμότητα. Και αυτό θα ήθελα να μου πει η Επιτροπή. Επιβεβαιώνει και αυτή η διαδικασία είναι πάντοτε ανοιχτή. Και δεν... Με ποια βάση παραμένουν ανοιχτέ. Δεν αφορά τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία, είτε είναι ορθή είτε μη ορθή. Διότι αυτό το οποίο ζητάει ο αναφέρον είναι ακριβώς αυτό έγινε μεταφορά νομοθεσία, αλλά εγώ δεν καλύπτομαι. Αυτό λέει. Ενώ άλλοι καλύπτονται, άλλο και εγώ. Και παρά το γεγονό ότι αυτή είναι μία αναφορά από ένα άτομο, θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με αυτόν. Γι' αυτό συμφωνώ ότι ένα άτομο μπορεί βεβαίως να προσφύγει στα εθνικά δικαστήρια. Αν όμως τέτοιες καταστάσεις πολλαπλασιαστούν και πολλά άτομα αντιμετωπίζουν τι ίδιε καταστάσει, τότε νομίζω πρέπει να το δούμε προσεκτικά, διότι ίσω υπάρχει δυσκολία στην ομοθεσία. Γι' αυτό παρακαλώ τον εκπρόσωπο τη Επιτροπή να μου δώσει συγκεκριμένε απαντήσει στα ερωτήματα. Ε, Σωστό. Ε, Μήπω πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί αυτή είναι η κεντρική ερώτηση, αν θέλετε. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο έχει φτάσει και στην Επιτροπή μα. Πολύ ωραία. Να, ξεκινήσω, να ξεκινήσω όμω με το γεγονό ότι εδώ υπάρχει μεγάλο βαθμό Μεγάλη σύγχυση. Πρέπει να σα εξηγήσουμε ότι η οδηγία δεν αφορά ένα αυτόματο δικαίωμα να έχει κανεί να μετατραπεί μια προσωρινή σύμβαση σε αορίστου χρόνου. Το οποίο σημαίνει ότι γι' αυτό ξεκινάνε πολλές αιτιάσεις, όχι μόνο στη Μάλτα, αλλά από την Ιταλία, τη Γαλλία, που οδήγησαν σε πολλές υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανέφερε σαφέστατα ότι τίποτε στην οδηγία δεν δίνει το δικαίωμα να μετατραπεί ε, το, η σύμβαση περιορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου. Και αυτό από εκεί ξεκινάμε. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μα. Αυτή είναι η αφετηρία. Το μόνο το οποίο κάνει η οδηγία είναι να προσπαθήσει να αποφύγει κατάχρηση ε, αυτή, αυτών των καταστάσεων. Που υπάρχουν δηλαδή συμβάσει ε, περιορισμένου χρόνου για πολλά χρόνια. Αλλά όταν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που δικαιολογούν αυτέ τι συμβάσει και δεν αντίκεινται στην οδηγία η αρχική παρατήρηση που βρίσκεται στη βάση αυτή τη διαδικασία ήταν η ε, παράπονο των γενικών γραμματέων των γραμματέων, όπου η νομοθεσία της Μάλτας που μεταφέρει την οδηγία δεν είχε προβλέψει κανένα μέτρο για να αποφευχθούν οι καταχρήσεις αυτών των κατηγοριών και ε, των τροποποιήσεων ε, που θα οδηγούν στη διαφοροποίηση μεταξύ αυτών των συμβάσεων και ώστε να μπορεί μια σύμβαση περισμένου χρόνου να γίνει ε, σύμβαση αορίστου χρόνου. Αυτό όμως συνέβη. Και αυτή, ε, αυτό αναφέρει η οδηγία η οποία βρίσκεται πίσω από το 2008, ότι πολλοί έχουν τακτοποιηθεί. Αλλά η οδηγία δεν εγγυάται, δεν δίνει εγγύηση, αυτόματη εγγύηση μετατροπής της προσωρινής σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Αυτό ίσως είναι το πρόβλημα. Το μόνο θέμα το οποίο παραμένει σε κρεμότητα αφορά τη διαγραφή ενός μικρού τμήματος των μέτρων μεταφοράς από τη Μάλτα που δεν έχουν καμία άμεση σχέση με ε, την αναφορά που βρίσκεται σε κρεμότητα. Και εκεί η Μάλτα πρόκειται να υιοθετήσει τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα ώστε να διαγραφεί αυτή η φράση in modifying. Και η Μαλτέζικη νομοθεσία όπως τροποποιήθηκε το 2008, διότι αυτό υπογραμμίζω πάντοτε, όπως τροποποιήθηκε το 2008, σύμφωνα με την Επιτροπή, είναι σύμφωνη με την οδηγία που αναφέρεται ε, στην μετατροπή των συμβάσεων περιορισμένης διαρκείας σε όριστη διαρκείας. Και είναι απόλυτα συμβατές με την οδηγία 9970. Ευχαριστώ κύριε have... Συγγνώμη, παίρνω και πάλι το λόγο, αλλά ε, ήθελα να γίνει αυτή η διευκρίνηση. Και με βάση αυτή την απάντηση τη Επιτροπή, θέλω να κάνω την εξή ερώτηση. Συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι Ορισμένοι τομείς, ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων έχουν εξαιρεθεί από την νομοθεσία της Μάλτας που μεταφέρει αυτήν την οδηγία σε εθνικό δίκαιο. Και πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το ότι έχουν εξαιρεθεί αυτές οι κατηγορίες είναι συμβατό με την οδηγία. Περί αυτού πρόκειται. Εδώ πρόκειται για κάποιο εκπαιδευτικό που είχε σύμβαση ορισμένου χρόνου που θεωρεί ότι έχει αποκλειστεί Έχουμε μια οδηγία που ισχύει για όλους τους εργαζομένους, γιατί επομένως να αποκλείεται κάποια κατηγορία, να αποκλείονται κάποιες κατηγορίες από τα ωφέλη της οδηγίας αυτής. Περί αυτού πρόκειται σε αυτή την αναφορά και γι' αυτό τώρα που αναδιατυπώνω το ερώτημά μου, πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει. Επιτροπή. Νομίζω ότι αρχικά το κύριο πρόβλημα με την ε, νομοθεσία αυτή που μεταφέρθηκε σε εθνικό δίκαιο ε, έχει καλυφθεί ε, μέχρι τώρα. Τα μέτρα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, τα μέτρα τα οποία θεσπίστηκαν δεν κάνουν, δεν κάνουν εξαιρέσεις για συγκεκριμένους τομείς. Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην νομοθεσία αφορούν ε, και τις συμβάσεις περιορισμένου χρόνου που πρέπει να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου και αναφέρεται και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που μπορεί να οδηγούν σε περιορισμένου χρόνου συμβάσεις. θα πρέπει επί 6-7 χρόνια να υπάρχουν συνεχείς συμβάσεις αορίστου χρόνου για να μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Όμως δεν εξαιρούνται κάποιοι τομείς. Ε, εφαρμόζεται αυτή η νομοθεσία για όλους τους τομείς, αλλά δεν δίνει αυτόματα δικαίωμα μετατροπής σε συμβάσεις αορίστου χρόνου είναι κάτι που το έχουμε δει και στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Νομίζουν οι πολίτες ότι μετά από 5, 6, 7 χρόνια αυτόματα μετατρέπονται οι συμβάσει ορισμένου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, αλλά δεν πρόκειται περί αυτού στην οδηγία. Δεν ξέρω αν ο συνάδελφος Μπουσούτη ε, καλύφθηκε. Ε, ακούσαμε ε, ότι η Επιτροπή πιστεύει ότι ε, συμφωνεί το θέμα αυτό με την ε, εθνική νομοθεσία η οποία ενσωμάτωσε την κοινοτική νομοθεσία. Εφιστά την προσοχή μας στο γεγονός ότι ε, όταν μιλάμε για μη ορθή εφαρμογή τη εθνική νομοθεσία, τότε αυτό δεν είναι δική μα αρμοδιότητα. Δεν ξέρω, κύριε Μπουσούτιλ, καλυφθήκατε, ε, κυρία Πρόεδρε, για να μην ε, σα καθυστερήσω άλλο. Θα ήθελα να τι κρατήσουμε ανοιχτές αυτές τις αναφορέ. Το παρακολουθώ και με την ώρα των επερωτήσεων στο Κοινοβούλιο. ήδη έχω αναφερθεί στο θέμα αυτό. Επαναλαμβάνω για μία τελευταία φορά. Αυτό που θέλω να πω εγώ δεν έχει να κάνει με το κατά πόσον η σύμβαση πρέπει να μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Αυτό είναι ένα πιθανό μέτρο που θα μπορούσαν να λάβουν ε, οι εθνικές αρχές και είναι δικό του ζήτημα. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι να δούμε κατά πόσον ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων μπορούν να εξαιρούνται από την εθνική νομοθεσία. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο, διότι η οδηγία δεν αποκλείει κάποια κατηγορία εργαζομένων. Δυστυχώς η, η, η απάντηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ικανοποιητική ω προ το σημείο αυτό. Γι' αυτό ζητώ να παραμείνουν ανοιχτέ οι αναφορέ αυτέ. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ε, με βάση το αίτημα του συνάδελφου Μπουσούτιλ μπορούμε να θεωρήσουμε, θα διατηρήσουμε ανοιχτή ε, και θα, την αναφορά αυτή και θα περιμένουμε συμπληρωματικές πληροφορίες για να καταλάβουμε κατά πόσον έχει δίκιο αναφέρον, ο οποίος μιλά για παραβίαση της κοινοτική νομοθεσίας. Δεν προκύπτει βέβαια κάτι τέτοιο με βάση τα δεδομένα και τα στοιχεία. Ε, ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή ε, ε, θα μπορούσε να μα δώσει κάποιε συμπληρωματικέ πληροφορίε. Γι' αυτό την κρατάμε ανοιχτή. Και τι δύο, και τις δύο ε, αναφορέ τι κρατάμε ανοιχτέ, περιμένουμε αυτέ τι συμπληρωματικέ πληροφορίε. Εάν συμφωνείτε, να πάμε στην επόμενη αναφορά. Στο σημείο 8, η 1287-2008 του Τζον Πάτρικ Για την αναφορά αυτή, νομίζω ότι όλα τα μέλη πήραν ένα συμπληρωματικό έγγραφο. Που και εγώ αυτή τη στιγμή το παίρνω το έγγραφο αυτό. Ο υπογράφων δεν είναι παρόν. που είχε πει ότι θα έρθει. Έστειλε όμως το έγγραφο γιατί δεν μπορούσε να έρθει. Να δώσω το λόγο λοιπόν στην κυρία Κανέτα Ρώση. Ευχαριστώ. Μια σύντομη ενημέρωση. Ίσως να πούμε και δύο λόγια για την ιστορία. Ο αναφέρον είναι πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος μετακόμισε στην Ισπανία και ε, καλύπτεται από το, ε, είναι ασφαλισμένο στο, ε, στο Ταμείο του Ηνωμένου Βασιλείου, έπαιρνε ένα ειδικό επίδομα βοήθεια που προβλέπεται για του Βρετανού υπήκοου από την Βρετανική νομοθεσία που χρειάζονται φροντίδα και τελικά δεν παίρνει πλέον το επίδομα αυτό, διότι οι αρχέ του Ηνωμένου Βασιλείου πιστεύουν ότι δεν πληρεί ένα από τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο για την παροχή αυτού του επιδόματος. Ε, αυτό το κριτήριο συνήθως το εξή. Από τις 52 ε, εβδομάδες ε, είναι παρόν μόνο τις 26 και ακριβώς για αυτό το λόγο του διεκόπη το επίδομα. Είναι παρόν στο Ηνωμένο Βασίλειο δηλαδή. Δεν βρισκόταν μάλλον τις 26 από τις τελευταίες 52 εβδομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο. η Επιτροπή εξέτασε την νομοθεσία που ε, ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση, ζήτησε πληροφορίες από, το, από τις αρχές του Ηνωμένου Βασίλειου, πήρε απάντηση ε, είδε ότι καλύπτεται από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του Ηνωμένου Βασιλείου ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ότι είναι ασφαλισμένος εκεί και μετά την ανάλυση καταλάβαμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Διότι θεωρούμε ε, ε, ότι αυτή, η, ότι αυτή προϋπόθεση να βρίσκεται στην επικράτεια του, της 26 52 εβδομάδας αντιβαίνει στην κοινωνική νομοθεσία. Και γι' αυτό το λόγο καταχωρήσαμε επίσημη καταγγελία κατά του Ηνωμένου Βασιλείου. Από το Σεπτέμβριο νομίζω, ε, σε αυτό το έγγραφο αναφέρεστε, ε, δώσαμε περαιτέρω πληροφορίε Σεπτέμβριο, λέγοντα ότι καταχωρήθηκε η αναφορά αυτή ω επίσημη καταγγελία. Τώρα, οι τελευταίε εξελίξει είναι εξή. Στι 9 Δεκάτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε ε, επίσημη ειδοποίηση ε, και ξεκίνησε τη διαδικασία παραβίασης κατά των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου ε, όσον αφορά αυτή την εθνική προϋπόθεση για τη χορήγηση του, του επιδόματος. Και δεν αφορά μόνο το επίδομα αυτό, αφορά και άλλα δύο επιδόματα. Δηλαδή τρία επιδόματα ομαδοποιούνται σε αυτή την περίπτωση και εκεί ισχύει ακριβώς η ίδια προϋπόθεση. Εμεί ε, ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούμε ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα και θέμα παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας. Ευχαριστούμε. Κύριε Γουόλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, δουλειά που έχουν κάνει. Και θα ήθελα να πω ότι από ό,τι φαίνεται δεν είναι μοναδική αυτή η αναφορά. Εγώ έχω πολλές περιπτώσεις ε, που ε, μου έχουν επισημανθεί από υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως επίσης και από οργανώσεις ατόμων με ειδικέ ανάγκες. Και είναι τεράστιο το πρόβλημα αυτό. Είναι πολύ δυσαρεστημένοι και δημιουργούνται προβλήματα σε πολλούς ανθρώπους από αυτή την ε, νομοθεσία και προτείνω το συντομότερο δυνατόν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Πριν από μια-δύο εβδομάδες λάβαμε μια σπαρακτική επιστολή από κάποιους πολίτες που ε, δεν είχαν λάβει τα επιδόματά τους και αυτό πραγματικά πρέπει να εξεταστεί. Και θέλω να σας παραπέμψω για κάποιες άλλες υποθέσεις για να τις εξετάσουμε από κοινού. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ και, και αυτή την αναφορά θα την αφήσουμε ανοιχτή περιμένοντας και περαιτέρω ε, πληροφορίε, λαμβάνοντα υπόψη και τι υποδείξει τη κυρία Γόλη. Μια απάντηση εκ μέρου του προσώπου τη Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Απλώς θέλω να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες, επιστολές, κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, οτιδήποτε μπορεί να απευθύνει κανείς προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και κυρίως αυτό το οποίο προσπαθούμε να επιτύχουμε είναι να μην δημιουργήσουμε εσφαλμένες προσδοκίες το κείμενο της Επιτροπής δεν μπορεί να σας βοηθήσει σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Αυτό είναι ένα θέμα που έχει σχέση με άτομα με αναπηρίες, με άτομα που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα και είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα, όπως είπε και η κυρία Wallis, και περιμένουν οι πολίτες που στέλνουν επιστολές συγκεκριμένες απαντήσεις. Εμείς εφαρμόζουμε την νομοθεσία και απλώς ε, εξηγούμε στους ενδιαφερομένους ότι βλέπουμε ποιο είναι το πρόβλημα, αλλά δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε και θα πρέπει σε εθνικό επίπεδο να το εξετάσουν. Ευχαρίστω λοιπόν να το εξετάσουμε όταν υπάρχει μια αναφορά, αλλά να έχουμε πάντοτε κατά νου ότι δεν πρέπει να γύρουμε ασφαλμένε προσδοκίε. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ε, ναι, έχετε δίκιο. Ε, λαμβάνω υπόψη αυτό που είπατε, να μην δημιουργούμε δηλαδή ε, αβάσιμες προσδοκίες. Αφήνουμε ανοιχτή λοιπόν και αυτή την αναφορά και πάμε στην επόμενη, στο σημείο 9. 590-2008 είναι παρόν αναφέρον. Noel Makulak. Καλησπέρα. Ευχαριστώ που με δέχεστε σήμερα εδώ. Για το θέμα αυτό της ε, αναφοράς μου υπάρχουν πολλά τα οποία έχουν προκύψει μεταξύ. Υπάρχουν ε, δύο σχετικά θέματα που αναφέρει η Επιτροπή ε, στην απάντησή της πέρυσι. Η νομολογία της Ιρλανδικής Δημοκρατίας, όπου αναφέρεται ότι γίνονται οι απαραίτητες αξιολογήσεις για την εφαρμογή της συνθήκης ε, Σέγγεν και έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά όχι για την Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Με λύπησε η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή για το θέμα αυτό. Ο κ. Έντουαρτ, σε μια επιστολή επικεφαλή της ε, μονάδας ε, πολιτικής ε, ουσιών, παρανόμων φαρμάκων, δηλαδή παρανόμων ουσιών και πιστεύω ότι δεν αντιμετωπίζονται τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με το δικό μου πρόβλημα των συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Φαίνεται σαν να έχω διαπράξει αξιόπινη πράξη και εγώ και άλλοι χρόνια ασθενείς ε, χρειαζόμαστε συνταγογραφούμενα φάρμακα και θα έπρεπε να ισχύει η αρχή ε, του ότι ε, θεωρούμε θα αθώοι μέχρι να αποδειχθεί οτιδήποτε διαφορετικό. Εγώ θέλω να έχω ελεύθερη κυκλοφορία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένη και τη Ιρλανδία. Και ε, αυτά τα οποία μου προσάπτονται είναι ε, ιδιαίτερα ε, επιβλαβή για μένα. Ήρθα σε επαφή το Μάιο του 2009 με το Κοινοβούλιο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα να, και να μπορώ να ταξιδέψω και στην Ιρλανδία. Ε, δυστυχώς στο αίτημά μου έλαβα την απάντηση ε, ότι δεν μπορούσαν να μου απαντήσουν άμεσα γιατί ήταν κλειστή μια υπηρεσία και έπρεπε να με παραπέμψουν σε μια άλλη υπηρεσία. Και ένας ε, υπάλληλος με ενημέρωσε ότι η καταγγελία της 13ης Ιουνίου θα έπρεπε ε, να απευθυνθεί στο δικό του τμήμα και όχι στο τμήμα ε, που ασχολείται με τα ναρκωτικά. Αυτά είναι τα ζητήματα με την Ιρλανδία και με την απάντηση του κ. Edwards. Και το Υπουργείο Υγείας στην Ιρλανδία το 2003 ενημέρωσε την Επιτροπή Ναρκωτικών των Ηνωμένων Εθνών, που είναι ο διεθνής οργανισμός που ασχολείται με το ψήφισμα 4415 των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μεταφορά φαρμάκων από ασθενείς για προσωπική χρήση, φάρμακα τα οποία περιλαμβάνουν και ψυχοτρόπες ουσίες, αλλά είναι συνταγογραφούμενα φάρμακα για αυτούς τους ασθενείς, και το Ιρλανδικό Υπουργείο ενημέρωσε την INCB, την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών δηλαδή, ότι θα πρέπει οι τελωνιακοί να αρκούνται σε μια επιστολή από το φαρμακείο ή από τον θεράποντα ιατρό που θα μιλά για την χρήση αυτών των φαρμάκων που βρίσκονται στην κατοχή του ασθενούς που ταξιδεύει. Στο πιστοποιητικό Σέγγεν όμως το Α, Β, Γ και Δ είναι πολύ διαφορετικές οι προποθέσει. Το πιστοποιητικό το οποίο προβλέπεται σύμφωνα με τη Συμφωνία Σέγγεν για τη μεταφορά φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών για προσωπική χρήση θα έπρεπε να παραπέμπει σε αυτά τα οποία ισχύουν και στα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα, όσον αφορά ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008, τον Οκτώβριο, μετά από μια εξέταση όλων των νομικών κειμένων, ε, κατέληξε στο ότι είναι δυνατόν να ταξιδεύει κανεί προ το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι νόμιμο αυτό με τα φάρμακα αυτά, αλλά όχι προ την Ιρλανδία. Το 2009 προσπάθησα να ασκήσω το δικαίωμά μου για ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν ήρθα σε επαφή με το Υπουργείο Εσωτερικών στο Ηνωμένο Βασίλειο με ενημέρωσαν ε, ότι υπάρχουν σχετικές διαδικασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τη μεταφορά φαρμάκων. Ήρθα σε επαφή με τον θεράποντα ιατρό μου και του ζήτησα να αλλάξει τη συνταγή και να μου δώσει Sativex, ένα φάρμακο το οποίο παρασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με την ε, σχετική νομοθεσία αν δεν άλλαζα το φάρμακό μου θα με συλλάμβαναν, θα μου κατέσχουν το φάρμακό μου και θα μου απίθυναν κατηγορία σαν να ήμουν ε, εγκληματίας. Το δικό μου φάρμακο ήταν το Bedrocan και το, βρετανικό, το φάρμακο του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν το Sativex, τα οποία είναι ταυτόσημα φάρμακα. Δεν βλέπω λοιπόν γιατί θα πρέπει εγώ να δίνω οδηγίες στον θεράποντα γιατρό μου να αλλάζει τη συνταγή φαρμάκων μου και εγώ δεν είμαι ιατρός ο ίδιος και δεν μπορώ να δίνω σχετικές ε, οδηγίες στην Ολλανδία. Δεν συνηθίζεται να δίδουν οι ιδιοκτικές αρχές ε, συνταγές ε, ασθενείς και θα πρέπει να γίνεται η απαραίτητη αξιολόγηση σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στην επιστολή του κυρίου Edwards από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις και δεν ε, προστατεύονται τα δικαιώματά μας. Κλείνοντα, θα ήθελα να πω ότι ε, είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα των χρονίων ασθενών και το Ηνωμένο Βασίλειο προσπαθεί να εμποδίσει χιλιάδες ε, ασθενείς ε, που έχουν προβλήματα με νόσους όπως το AIDS, η ή οτιδήποτε άλλο και προσπαθεί να του εμποδίσει από το να μετακινούνται στην Αγγλία και στο Λονδίνο ενώπιση και των Ολυμπιακών του 2012. Με βάση τις ε, τρέχουσες ιατρικές γνώσεις για την διατήρηση της υγείας μας, θα πρέπει ε, να έχουμε μια ελπίδα για βελτίωση της κατάστασής μας, ιδιαίτερα για τους ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο. Σε ασθένειες όπως η σκλήνση κατά πλάκας υπάρχουν φάρμακα τα οποία βοηθούν. Υπάρχει ε, το τεσάμπλ στην Ιρλανδία που εξάγεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ιρλανδία, αλλά υπάρχει ε, ο κίνδυνος θανάτου, ακόμη και ε, ένα στις 600 περιπτώσεις να είναι, ε, ο κίνδυνος θανάτου ως παρενέργεια για μένα είναι αποτρεπτικός. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και σας εύχομαι καλές γιορτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και αν βρίσκεστε και εσείς και η οικογένεια σας. Εγώ σας ευχαριστώ να δώσουμε το λόγο στην κυρία Μαρή Ντεμπίβ εξ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι εδώ. Όχι, όχι, λάθος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώς να διευκρινίσω το εξή. Δυστυχώ η Μαρή βεβαίω, η οποία είναι ο δικηγόρο στη μονάδα μας, δεν είναι εδώ, ζητώ συγγνώμη, έγινε μια μικρή παρεξήγηση λόγω του ονόματο τη μονάδα μα που ονομάζεται Anti-Drugs Unit. Αλλά έτσι ονομάζεται, δεν φταίμε εμείς, ο ρόλος όμως της μονάδας μας είναι να συντονίζει όλες τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με τα φάρμακα ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό δεν υποτίθεται ότι κάποιος είναι εγκληματίας τη στιγμή, δεν είναι κατά των ναρκωτικών. Δεν ε, ασχολούμαστε με τα θέματα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Επειδή είμαστε Επιτροπή, έχουμε ε, διαβουλευτεί με τους υπεύθυνου του Σέγγεν, με εκείνους που ασχολούνται με την ελεύθερη διακίνηση. Συνεπώς, ζητώ συγγνώμη, εάν αυτό δημιούργησε προβλήματα ή κατά πόσο αυτό ήταν παραπλανητικό ως προς τη φύση της μονάδας μας. Καταλαβαίνω αυτά τα οποία ε, σας έγραψε ο κ. επικεφαλής μονάδος και υπάρχουν όλες οι νομικές λεπτομέρειες που δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Η Μαρία από τη μονάδα μας, η οποία είναι νομικός, ε, θα ασχοληθεί με τις νομικές λεπτομέρειες. Εγώ με τα χαράς είτε να απαντήσω σε ερωτήματα που έχετε εκτός του νομικού πλαισίου, εδώ ή κατηδίαν. Αλλά θα δώσω το λόγο τώρα στη Μαρία να σας απαντήσει για τα νομικά θέματα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καταστήσω σαφές το εξής. Το Ιρλανδικό πρόβλημα και το Βρετανικό πρόβλημα είναι δύο θέματα. Εμείς ε, λάβαμε την επιστολή σας σχετικά με το πρόβλημα που έχετε με την πωλήση των εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από δύο εβδομάδες. Υπάρχει νομίζω παρεξήγηση. Ο κύριος Έντουαρτς ε, στην επιστολή του του 2008 αναφερόταν στην Ιρλανδική περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν το πρόβλημα ήταν ότι το άρθρο 75 της ε, Συμφωνίας Εφαρμογής του Σέγγεν δεν καλύπτει ε, τους ε, ταξιδιώτες που έχουν ε, φάρμακα και η Ιρλανδία ζήτησε να περιληφθεί σε αυτή τη συμφωνία. Αλλά η απόφαση του Συμβουλίου του 2002 Και αλλά η εφαρμογή αυτών των διατάξεων του άρθρου 75 εξαρτάται από μία άλλη απόφαση του Συμβουλίου, η οποία δεν έχει ληφθεί υπόψη. Legal point. Γι' αυτό από καθαρά νομική άποψη, αυτό το άρθρο δεν είναι δεσμευτικό για την Ιρλανδία. Συνεπώς, ε, δεν σημαίνει ότι υπάρχει παραβίαση της κοινωνικής νομοθεσίας από την Ιρλανδία. Για την Ιρλανδία, τώρα για το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είπατε πριν από δύο εβδομάδες, γνωρίζομαι ότι είχατε, σχέση, ότι είχατε σε επαφή με το Υπουργείο Ιστορικών και η νομική υπηρεσία ε, του Υπουργείου Ιστορικών ασχολείται με την υπόθεση και προσπαθεί να δει πού βρίσκεται αυτό το θέμα και εμείς παρακολουθούμε το θέμα για να δούμε πώς εφαρμόζουν το άρθρο 75. Στη δική του την περίπτωση είναι δεσμευτικό τα δύο θέματα λοιπόν της Βρετανίας και της Ισλανδίας είναι εντελώς διαφορετικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μία ε, υπόθεση που πραγματικά είναι στο επίπεδο ε, των ε, όσων διαβάζουμε στον Κάφκα. η πλήρη νίκη τη γραφειοκρατίας κατά των Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με εγκληματίε. Δεν έχουμε να κάνουμε με άτομα που προσπαθούν να μεταφέρουν ναρκωτικά. Μιλάμε για ένα Ευρωπαίο πολίτη που θέλει να γυρίσει στη χώρα του, είτε για να ψηφίσει, είτε γιατί θέλει να επισκεφθεί τη χώρα του, για οποιοδήποτε λόγο. Και δεν του επιτρέπεται γιατί δεν υπάρχουν οι σχετικέ νομικές διατάξεις ή γιατί δίνεται ιδιαίτερα γραφειοκρατική ερμηνεία της νομοθεσία και δεν επιτρέπεται στον συγκεκριμένο πολίτη να υποφεληθεί των δικαιωμάτων του. Τεχνικά είναι σωστές οι πληροφορίε της Επιτροπής. Αλλά ω μέλος της επιτροπή Αναφορών και ως Ευρωπαίος πολίτη. Θέτω το ερώτημα αν όντω έχουμε το δικαίωμα να θέτουμε σε κίνδυνο τη ζωή ενός πολίτη με αυτά τα γραφειοκρατικά μέτρα. Δεν μπορεί οι διοκτικέ αρχές να αλλάζουν τα φάρμακα που συνταγογραφούνται σε έναν ασθενή και στη χώρα μου, στη Ρουμανία, θα ήταν εγκληματική ενέργεια κάτι τέτοιο δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση από ό,τι γνωρίζουμε, αλλά τι να πούμε στους πολίτες της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν μια τέτοια κατάσταση. Πιστεύω ότι είναι επίγον το θέμα και έχουμε αρμοδιότητες τις οποίες δεν μπορούμε να παραβλέψουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι απλώς περιμένουμε μια απάντηση από την Ιρλανδική ή την Βρετανική κυβέρνηση. Πρόκειται για εντελώς παράλογη κατάσταση. Δεν λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα των πολιτών μας. Είναι απαράδεκτο αυτό και πρέπει να αλλάξει άμεσα. Διαφορετικά δεν μπορούμε να αποκαλούμε θα Ευρωπαϊκή Ένωση Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό αυτή την έννοια είναι θύμα πρακτικών που πρέπει άμεσα να αλλάξουν. Δεν είμαι νομικός. Και δεν έχω απάντηση να δώσω σε έναν πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζει μια τόσο δύσκολη κατάσταση. αποτελεί αποτυχία των εθνικών και των ευρωπαϊκών αρχών αυτή η κατάσταση. Οι πολίτες θέλουν να χαίρουν των δικαιωμάτων τους. Äh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συμφωνήσω κι εγώ με τα λεγόμενα του προηγούμενου ομιλητού, αλλά εδώ έχουμε ένα ε, ε, βασικό πρόβλημα. Εμείς ως Επιτροπή Αναφορών λαμβάνουμε αναφορές σε ορισμένες περιπτώσεις είναι μη παραδεκτές ε, οι αναφορές. Εδώ καταλαβαίνουμε εμείς ότι ο αναφέρον έχει δίκιο και πρέπει να τον βοηθήσουμε για ανθρωπιστικούς λόγους. Από την άλλη πλευρά ακούμε και τα τεχνικά επιχειρήματα της, Επιτρο... της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ακούμε ποιο είναι το ισχύον δίκαιο. Μπορεί να είναι, ε, να μην πω απάνθρωποι, αλλά ε, να είναι μια ε, νομική απάντηση που δεν μας καλύπτει για αυτό το οποίο θα θέλαμε για ανθρωπιστικούς λόγους να εφαρμόσουμε εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε μέτρα, να κάνουμε κάτι και να, να φροντίσουμε να αλλάξει κάτι όταν η νομική αντιμετώπιση είναι απάνθρωπη. Τι κάνουμε, τουλάχιστον να στείλουμε μια επιστολή προς την Επιτροπή. Εμείς συμφωνούμε ότι δεν μπορεί να παραμείνει έτσι η κατάσταση. Είναι μη ικανοποιητική αυτή η κατάσταση, αν μα λένε ότι από τεχνική ε, άποψη αυτή έχει η κατάσταση. Εμεί καθόμαστε εδώ ω ευρωβουλευτέ ε, σήμερα και όλε που τίθεται σε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνα. Δεν μπορούμε να μην κάνουμε τίποτα. Γιατί είναι τελώς παράλογη αυτή η κατάσταση. Να μην μπορούμε να βοηθήσουμε έναν αναφέροντα γιατί υπάρχει μια αντίθετη νομική βάση. Πρέπει οπωσδήποτε ε, να γίνει κάτι. Ε, υπάρχουν ε, πάρα πολλοί ασθενείς που έχουν συνταγές από το θεράποντα ιατρό τους σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παίρνουν τα φάρμακά τους μαζί στο αεροπλάνο και πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν και όχι να τους περιορίζεται η πρόσβαση σε μια άλλη χώρα γιατί το συγκεκριμένο φάρμακο μπορεί να θεωρείται ναρκωτική ουσία. Εμεί ω Επιτροπή Αναφορών ε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Ε, Ευχαριστώ. Ο κύριο Άτκιν έχει το λόγο. Α, η κυρία. Ε, σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στο συγγνώμη που δεν ήμουν στην αρχή τη παρουσίαση, αλλά συμφωνώ και με του δύο από του τελευταίου ομιλητέ και να μην επαναλάβω αυτό το οποίο είπαν. Νομίζω ότι εδώ το ζήτημα ε, ανάγεται στο εξή. Τι μπορούμε να κάνουμε ω Επιτροπή Αναφορών εμεί. Μία από τις ε, δηλώσει τη Επιτροπής στην απάντησή τη ήταν ότι η απόφαση δεν έγινε σε σχέση με την Ιρλανδία γιατί δεν έχει γίνει ακόμα η σχετική αξιολόγηση, μα έχει γίνει. Ε, όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο. Και βεβαίω στη συνέχεια αναφέρει παρακάτω ότι ένα από του λόγου ενδεχομένως γιατί δεν έγινε είναι ε, ε, λόγω του ότι η Ιρλανδία θέλει αναβολή έτσι ώστε να συνδεθεί με τη δεύτερη γενιά του πληροφοριακού συστήματο Σέγγεν που αναμένεται να είναι λειτουργικό μέχρι το τέλο του 2009. Έχω λοιπόν ερώτηση προ την Επιτροπή. Αν αναμένεται να είναι λειτουργικό μέχρι το τέλο του 2009 Μπορούμε εμεί τώρα, γιατί είμαστε στο τέλο του 2009, μπορούμε ε, ε, μπορεί να γίνει με ταχύτητα η αξιολόγηση και να προχωρήσουμε με, βάση από τη νομική του σκοπιά. Καταλαβαίνω αυτό που είπαν οι προλαλήσαντες και ακούγοντα και τον αναφέροντα και, και άκουσα και την κατάστασή του. Αλλά η θέση μα είναι εξή. εμεί τι μπορούμε να κάνουμε με νόμιμο τρόπο, από νομική άποψη, για να προωθήσουμε το ζήτημα. Ίσως λοιπόν θα μπορούσε να ξεκαθαρίσει το ζήτημα η Επιτροπή με την αξιολόγηση, να δούμε τον αντίκτυπο στη συνολική κατάσταση και να δούμε αν υπάρχει κάποιο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε ε, ότι αυτό θα γίνει γρήγορα και στη συνέχεια να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Ή μήπω υπάρχουν άλλα μέτρα τα οποία θα μπορούσαμε να λάβουμε για παράδειγμα, ο αναφέρον ε, έχει και μία καταγγελία σε σχέση με το γεγονό ότι ε, το Ιρλανδικό Υπουργείο Δικαιοσύνη δημοσίευσε τα, ε, τα ιατρικά του δεδομένα. δεν θα μπορούσαμε και εδώ να κάνουμε κάτι. Το αφήνω όμω σε εσά, Πρόεδρε, το ζήτημα. Ευχαριστώ. Higgins. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αυτή η οδηγία ή αυτή η απόφαση του Συμβουλίου είναι το 2002, δηλαδή πριν από 7 χρόνια. Προς τι να μιλάμε για την υποστήριξη των δικαιωμάτων πολιτών όταν μόνο στο χαρτί υπάρχουν και όχι στην πράξη. Η έκθεση λέει το άρθρο 4 αναφέρει ότι θα πρέπει το άρθρο 1 να εφαρμοστεί, αλλά η απόφαση του Συμβουλίου δεν αναφέρει προθεσμίες. Συνεπώς, Πού βρισκόμαστε εμείς από πλευρά αναφέροντος. Και θα σας πω ότι αυτό αφορά και τους πολίτες της Ιρλανδίας που διαμένουν στην Ιρλανδία και έχουν κάποια ασθένεια. και θα μπορούσε αυτό το φάρμακο να τους ανακουφίσει. Η Ιρλανδική κυβέρνηση δεν θέλει να το βλέπει αυτό το θέμα διότι πληρώνουμε πάρα πολλά χρήματα σε πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες για συνθετικά φάρμακα, αλλά κάτι το απλό, το οποίο μπορεί να ανακουφίσει τόσο κόσμο και σε σωστές συνθήκες απαγορεύεται παντελώς. Νομίζω λοιπόν ότι η Επιτροπή θα πρέπει να το διευκρινίσει. Δηλαδή να μας πει πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η διάταξη και τι μπορεί να γίνει ώστε να μπορούμε να οθήσουμε και την ελληνική κυβέρνηση να το κάνει. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να προσθέσει ή να ξεκαθαρίσει κάτι, αν το επιθυμείτε βεβαίως. Sí. On, on the λοιπόν, για το θέμα της Ιρλανδίας. Αυτή η επιστολή είχε συνταχθεί πριν από ένα χρόνο, όταν είχαμε σκεφτεί ότι θα είχε εφαρμοστεί στο τέλος του 2009. Προφανώς είχα επαφές με τη μονάδα Σέγγεν, διότι εμεί δεν ασχολούμεθα απευθεία με αυτό το θέμα. Τίποτα δεν άλλαξε δυστυχώς. Αλλά είναι επίσης προφανές ότι δεν αναπόκειται στην Επιτροπή να οθήσει να σπρώξει την Ιρλανδική κυβέρνηση. Εμείς δώσαμε αυτές τις πληροφορίες που είχαν σχέση με αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν φαίνεται ότι η κυβέρνηση της Ιρλανδίας να θέλει να εφαρμόσει τώρα αυτή τη διάταξη. Συνεπώς αυτό είναι ένα θέμα εθνικής πολιτικής. I would like to ask the Commission a very straight... Σας παρακαλώ, θέλω να κάνω μια ερώτηση ξεκάθαρη προς την Επιτροπή, για να μην ε, έτσι ε, ξεφεύγουμε σήμερα το απόγευμα και ξελιστράμε, για να ρωτήσουμε. Έχουν ξεκινήσει διαδικασίε παραβίαση κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Δύο εβδομάδε όταν πήρατε την επιστολή αυτή και το ελέγξατε του συναδέλφου σα ε, που είναι υπεύθυνοι στο Υπουργείο Δικαιοσύνη. Περιμένουμε ε, έχουμε ζητήσει πληροφορίε από το Υπουργείο Δικαιοσύνη. Τα Χριστούγεννα είναι στι δύο-τρει εβδομάδε. Γιορτή τη Χριστιανοσύνη. Έχω χάσει τρει φορέ τα Χριστούγεννα. Αν ξέρετε, πριν από λίγο καιρό ε, η πατρίδα μου, ε, το χωριό μου, πλημμύρισε. Άρα μπορεί να μην έχω καν χωριό να επιστρέψω με την, από αψιουσία, αλλά ίσω μπορούσα να, να επιστρέψω και εγώ να τη βοηθήσω στην νοικοδόμηση. Λοιπόν, κοιτάξτε, με βάση αυτά τα οποία ακούσαμε από την Επιτροπή, και με τις παρεμβάσεις των συναδέλφων, εμείς ως Επιτροπή Αναφορών αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα να αποστείλουμε ένα σημείωμα προς τις Εθνικές αρχές. να τονίσουμε τη, την ε, δυσφορία μας και, να ζητήσουμε να ληφθεί απόφαση και σε σχέση με αυτά τα οποία ε, αναφέρθηκαν ο συναδέλφος Χίγκινς. Όσον αφορά δηλαδή ε, το χρονοδιάγραμμα και το τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ε, νομίζω ότι εμείς ως Επιτροπή Μεταφορών, Αναφορών συγγνώμη, μπορούμε να ζητήσουμε επιγόντως να δοθεί μια απάντηση από τις εθνικές αρχές. Τουλάχιστον εν μέρη να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια απάντηση ε, στον αναφέροντα. Ε, ας προσπαθήσουμε λοιπόν να δώσουμε μια απάντηση. Τα Συμφωνείτε ε, να θεωρήσουμε λοιπόν εμεί ω Προεδρία ότι μπορούμε να αποστείλουμε μια, ένα σημείωμα προ τι Εθνικέ Αρχέ. Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και τον αναφέρω. Πάμε στο 10. 1688-2008, George Mills, με ε, παρόντα των υπογραφών, τον οποίο και δίνουμε το λόγο. Uh, Το απόγευμα, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που μας επιτρέπετε να δώσουμε συνέχεια σε αυτή την αναφορά. Τα πράγματα λίγο προχώρησαν από τότε που κατατέθηκε η αναφορά και θα σας δώσω το γενικό ιστορικό. Προφανώς ο αναφέρον είναι κατά της μεμονωμένης καταγραφής και της ηλεκτρονικής επισήμανσης στα εγώ πρόβατα. Και αυτό το θέμα είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε, ώστε να δούμε πώς ε, γίνονται οι καταγραφές. 8.000 ε, και περισσότερα άτομα έχουν υπογράψει αυτή την αναφορά μόνο από τη Σκοτία. Από τότε τα πράγματα έχουν προχωρήσει και άλλες χώρες γνωρίζουν πλέον το πρόβλημα το οποίο θα υπάρξει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και μάλιστα τώρα υπάρχουν 14 χώρες που έχουν αναφέρει ότι υπάρχουν προβλήματα για τον ΑΒ λόγο με αυτό το σύστημα. Αλλά το πραγματικό πρόβλημα εδώ είναι ότι αυτές οι 14 χώρες αντιπροσωπεύουν 60 εκατομμύρια και περισσότερα εγωπρόβατα. Δηλαδή πάνω από το 50% των συνολικών εγωπροβάτων στην Ευρώπη. Τα πράγματα λοιπόν έχουν πολύ προχωρήσει από την εποχή που είχε κατατεθεί η πρώτη αναφορά. Και ο λόγος, ο πραγματικός λόγος, είναι ότι τα εγωπρόβατα είναι ουσιαστική σημασία για την αγροτική οικονομία στη χώρα μας. Για να σας δώσω μια ιδέα σχετικά με τα στοιχεία της σκοτίας μόνον, 170 εκατομμύρια ε, κεφάλια υπάρχουν ε, πρόβατα στη σκοτία και όχι μόνο ω εισόδημα, αλλά αυτό έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην αγροτική ε, οικονομία και συνεπώς δημιουργείται μία λίρα ε, επιπλέον για την οικονομία. Αν το πολλαπλασιάσετε σε όλη την Ευρώπη, βλέπετε ότι μιλάμε για πολύ σημαντικούς αριθμούς και για ένα σημαντικό κεφάλαιο των αποπροβάτων για την ευρωπαϊκή οικονομία. Και όχι μόνο αυτό υποστηρίζει την αγροτική οικονομία και την οικονομία γενικά, αλλά και το περιβάλλον, διότι αναπτύσσεται και ο τουρισμός. Αυτό που μας απασχολεί λοιπόν είναι να σταματήσει αυτή η καταγραφή ε, των εγωπροβάτων, να ξαναδούμε αυτό το θέμα και τώρα θα δώσω ε, το λόγο στο συνάδελφό μου, τον κύριο Μίλνα. Ευχαριστώ. Αναγνωρίζετε ότι 30 μέρες πριν από την εφαρμογή του κανονισμού, ο κλάδος μας θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το επιπλέον βάρος. Νομίζω όμως ότι ε, ο προβληματισμός σε όλη την Ευρώπη έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι διαβουλεύσεις ε, για τους νέους κανονισμούς ε, για την υγεία των ζώων του 2007 αφορά και την σήμανση των ζώων. Και αυτό αποτελεί μέρος των διαβουλεύσεων. Και αναφέρω ότι αυτά τα μέτρα θα έχουν πολλά ωφέλη για, σε πολλούς τομείς. Αλλά αυτοί οι σημερινοί κανόνες υπογραμμίζουν περισσότερο τις τεχνικές λεπτομέρειες παρά τις αρχές και τους στόχους. Συνεπώς, για ορισμένους ενδιαφερόμενους ήταν δύσκολο να του δεχτούν. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί εάν υπάρχει πιο συνεκτική και πιο απλή νομοθεσία. Γι' αυτό παρακαλούμε την Επιτροπή σας και τους ε, ευρωβουλευτές να διευκολύνουν την αθεώρηση του κανονισμού 21-2004, λαμβάνοντας υπόψη ε, τον προβληματισμό των ενδιαφερομένων. Και να υπάρξει μια πιο στοχοθετημένη εφαρμογή ε, που θα είναι καλύτερη για, την, για τον κλάδο μας. Ευχαριστώ. Αυτό είναι το έτοιμά μας. Αυτή είναι... Ευχαριστώ. Το λόγο έχει Επιτροπή. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο κανονισμός που ανέφεραν οι αναφέροντες 21-2004 υιοθετήθηκε το 2003 μετά από την επιδημία του φόδου πυρετού και κυρίως μετά από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω των εκθέσεών του σχετικά με τον αυθόδη πυρετό. Και όχι μόνο μετά από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και του ελεγκτικού συνεδρίου και άλλων εθνικών εκθέσεων. Αυτές οι εκθέσεις είχαν ως αντικείμενο να ενισχύσουν τους κανόνες ιχνηλασιμότητας για τα εγωπρόβατα, όπου υπήρχε μεγάλη εξάπλωση του φθόδου σπυρετού στον Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και σε άλλες χώρες. Συνεπώς, η Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο πρότασης που παρουσίαζε διάφορα μέτρα ιχνηλασιμότητας, ατομικής ιχνηλασιμότητας και ηλεκτρονικής αναγνώρισης για τα εγωπρόβατα. Αυτό εισήχθη βαθμιαία και το 2007 το Συμβούλιο όρισε την ημερομηνία για την ηλεκτρονική καταγραφή των αγοπροβάτων, δηλαδή την 31η Δεκεμβρίου 2009. Το Συμβούλιο όμως δεν ακολούθησε την αρχική πρόταση της Επιτροπής η οποία έλεγε ότι θα πρέπει αυτή η ημερομηνία να καθοριστεί μέσω της επιτροπολογίας. Αλλά το Συμβούλιο ακολούθησε την ε, νομοθετική, το νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όρισε την ημερομηνία στην 31η Δεκεμβρίου 2009. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή προσπάθησε να διευκολύνει την ομαλή εισαγωγή της ηλεκτρονικής καταγραφής των εγωπροβάτων και ε, το παράρτημα μέσω της Επιτροπολογίας και η Επιτροπή ξεκίνησε μία μελέτη ε, του Κοινού Κέντρου Ερευνών για ε, την οικονομική ανάλυση των διαφόρων επιλογών για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής αναγνώρισης και η Επιτροπή παρακολούθησε ε, τις συζητήσεις που έγιναν στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα και κυρίως ε, τις προτάσεις ε, που έγιναν από τους ευρωβουλευτές και την έκθεση για την κατάσταση που βρίσκεται το τομέα των εγωπροβάτων τους. Επίσης, τις συζητήσεις στο Συμβούλιο Γεωργίας τρεις φορές φέτος πολλά κράτη-μέλη έθιξαν αυτό το θέμα στα διάφορα. Αλλά στο Συμβούλιο δεν δόθηκε ποτέ ένα σαφές μήνυμα ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα ήθελαν να αλλάξουν αυτή την αρχή της ατομικής συχνηλασιμότητας των εγωπροβάτων. Και συνεπώς η κατάσταση είναι ακριβώς αυτή που σας περιέγραψα. Ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο στο συνάδελφο Σμιτ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να υποστηρίξω την αναφορά αυτή, όπως ε, έκανα και όταν ήρθε εδώ στην Επιτροπή μας, γιατί είναι ευρωπαϊκό ζήτημα και τότε ήταν και τώρα. Δεν αφορά μόνο ε, την, ε, τη, σήμανση, αλλά αφορά την καλύτερη νομοθέτηση. Και με αυτή την έννοια μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ε, γιατί πραγματικά εδώ μιλάμε για νομοθεσία που έχει μαζικές επιπτώσεις στον πραγματικό κόσμο και να δούμε και να δείξουμε τι γίνεται ε, όταν ακριβώς ε, αποφασίζει την νομοθεσία αυτή. Πρέπει να σας πω ότι ε, πραγματικά έγιναν αλλαγές στον κανονισμό από τότε που ήρθε η αναφορά ε, και βεβαίω είναι καλέ οι αλλαγέ. Αναφέρθηκε ήδη ότι συζητήθηκε τρει φορέ στο Συμβούλιο Γεωργία το ζήτημα. Τρει φορέ, Όχι γιατί είναι, υπάρχει κάποιο που να είναι ικανοποιημένο, αλλά επειδή όλο και περισσότερα κράτη-μέλη δεν είναι ικανοποιημένα με τι διατάξει του πακέτου. Και ειλικρινά απογοητεύομαι ε, γιατί ε, πολλοί καθυστέρησαν να καταλάβουν ποιε είναι οι πραγματικέ επιπτώσει όλων αυτών. Πάντω υπήρξε μεγάλη ανησυχία όσον αφορά τι επιπτώσει. Σε αυτού του νομοθετικού πακέτου. 14 κράτη-μέλη τώρα υποστηρίζουν το γεγονό ότι υπάρχουν πρακτικά προβλήματα, υποστηρίζουν την άποψη αυτή και εξακολουθούμε να είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι για τι επιπτώσει στον τομέα τη κτηνοτροφία. Από άψη κόστου, από άποψη ε, ε, μειωμένη ε, ασφάλεια εφοδιασμού στον τομέα των τροφίμων και μάλιστα σε μια εποχή όπου θα έπρεπε να κάνουμε ε, τα πάντα για να, για να προωθήσουμε τον κλάδο. 30 ημέρε μα χωρίζουν από την ε, υλοποίηση και την εφαρμογή του κανονισμού, το καταλαβαίνουμε Χαιρόμαστε που υπήρξαν αλλαγέ, αλλά εξακολουθούμε να ανησυχούμε ιδιαίτερα γιατί πιστεύουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πρακτικέ δυσκολίε όσον αφορά την εφαρμογή τη πρόταση και του κανονισμού. Και προτείνω ε, το, θέμα αυτό να εξακολουθήσουμε να, να θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να και, πραγματικά ε, να προχωρήσουμε προς την αλλαγή της νομοθεσίας υπό τον δημοκρατικό έλεγχο του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας. 14 κράτη-μέλη εξέφρασαν επιφυλάξεις απέναντι σε αυτό το πακέτο. Ε, συμφωνήθηκε πριν από αρκετό καιρό όταν υπήρχαν διάφορες προσδοκίες σε σχέση με την τεχνολογία όπου δεν πρόσεξαν ιδιαίτερα. Άρα λοιπόν τέλος πάντων δεν έχουμε σημασία όλα αυτά. Πρέπει να τα διορθώσουμε και να διορθώσουμε ε, την νομοθεσία. Ε, στα πλαίσια της βελτιωμένης νομοθεσίας είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατήσουμε το θέμα επίκαιρο ε, στην ε, ημερήσια διάταξη, στο επίκεντρο τη σκέψη μα και του προβληματισμού μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Τσίτσεστερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να μιλήσω ε, υποστηρίζοντας τους αναφέροντες. Εκπροσωπώ ένα διαφορετικό, ε, μια διαφορετική περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην άλλη άκρη ε, σε σχέση με τη Σκωτία. Αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν ευρύτερες ανησυχίες όσον αφορά την επίπτωση του μέτρου αυτού. Ευρύτερη ανησυχία ε, στον κλάδο της κτηνοτροφίας και στους γεωργούς Ακριβώς γιατί υπάρχουν ορισμένα πρακτικά στοιχεία που αφορούν την υλοποίηση και την εφαρμογή, όπως είπε και ο συνάδελφος. Νομίζω ότι ε, είναι... Ε, κοιτάξτε, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στο γεγονό ότι ποτέ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαφώνησε με τον κανονισμό. είναι κάπω υπερβολικό αυτό το οποίο λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εάν είχαμε εδώ τον αμέσω προηγούμενο πρόεδρο τη Επιτροπή Γεωργίας, θα διαφωνούσε ιδιαίτερα. Θα το κάνω εγώ για λογαριασμό του συναδέλφου. Και νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει ε, ε, να ντρεπόμαστε απέναντι σε λάθος, ε, απέναντι σε τέτοια ε, παραπληροφόρηση και, ε, λάθος, απέναντι σε τέτοιε ε, λάθος αναφορές. Ξέρω, παρόλο που δεν είμαι ειδικό, ότι υπάρχουν πολλέ πρακτικέ δυσκολίε. Θυμάμαι πριν από ορισμένα χρόνια, σε μία επίσκεψή μου, ε, είδα εκεί ε, τα, τα συστήματα ηλεκτρονικού εντοπισμού ε, και μου τα έδειχναν εκεί οι ειδικοί με, με υπερηφάνεια. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αποδείξει ότι είναι σωστά όλα αυτά. Αλλά δεν πιστεύω εγώ ότι με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε τις νόσους. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει περαιτέρω ε, ε, αξιολόγηση αντικτύπου, ανεξάρτητη και όχι που να βγαίνει από τις έπες της και, να την, και υπό την επίβλεψη του Κοινοβουλίου. Υποστηρίζω απόλυτα αυτά που ο συνάδελφο, λοιπόν κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Λάιον έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Και εγώ ως νέο μέλος θα ήθελα να υποστηρίξω την αναφορά την οποία έχουμε εδώ, εδώ και το καιρό. Και όπως είπε και ο συνάδελφος Σμίθ και ο κύριος Τσίσοστε, που επίσης μίλησαν υπέρ ε, της αναφοράς, θα ήθελα και εγώ ε, να δω την αναθεώρηση του κανονισμού και κυρίως όσον αφορά τις πρακτικές επιπτώσεις. Πιστεύω ότι η πρακτική, το πρακτικό αποτέλεσμα του κανονισμού είναι δυσανάλογο με τους στόχους Επιτροπής να υπάρχει ένα λογικό σύστημα εθνηλασιμότητας για να είναι βέβαιο ότι υπάρχει προστασία των ζώων από τις ασθένειες. Και γι' αυτό ε, θα ήθελα η αναθεώρηση να εστιάζεται στην ανάγκη της καταγραφής των εγωπροβάτων που δεν ε, κυκλοφορούν μακριά από το κτήμα μέχρι την ημέρα της φαγής τους. Λοιπόν, θα πρέπει ο κάθε κτηνοτρόφος να το ξέρει, διότι τα εγωπρόβατα για 5 ή 6 χρόνια δεν μετακινούνται και τότε θα πρέπει οι κτηνοτρόφοι να εγγυώνται την καλή κατάστασή τους. Επίσης, θα πρέπει να θεωρήσει να δει ε, κατά πόσον τα λιγότερα μέτρα, λιγότερα μέτρα ε, θα μπορούσαν να ληφθούν όπως έχουμε στη Σκωτία, στη Βόρεια Αγγλία και στην Ιρλανδία. Αλλά επίσης πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένα δίκαιο παιχνίδι σε όλη την Ευρώπη ω προ την εφαρμογή των μέτρων. Και μου επιβεβαιώθηκε ότι η Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα χρηματοδοτούν τους κτηνοτρόφους μέσω των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης για να μπορέσουν να εφαρμόσουν τη νέα τεχνολογία και τα νέα συστήματα και κυρίως ε, βοηθάνε τις μονάδες, τις χρονοτροφικές μονάδες. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει το παιχνίδι να είναι δίκαιο όσον αφορά τη χρηματοδότηση, ε, διότι η κυβέρνησή μας του Ηνωμένου Βασιλείου και της ε, Ιρλανδίας θα πρέπει να χρηματοδοτεί επίσης τους χρονοτρόφους. Επίσης πρέπει να δούμε κατά πόσον αυτός ο κανονισμός είναι ανάλογος ή δυσανάλογος. Η Επιτροπή δεν μου Δηλαδή ότι δεν θα, υπάρχουν, δεν θα χρειάζεται εισαγωγέ από τρίτες χώρες να έχουν το ίδιο επίπεδο ειχνηλασιμότητα στι χώρες τους. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το λύσουμε. Θα πρέπει πάλι και εδώ το παιχνίδι να είναι ισότιμο, να είναι δίκαιο για όλους όσους ε, ασχολούνται με την κτηνοτροφία εγώ προβάτων και έχουν ε, εισαγωγές των ζώων από άλλε χώρε. Ο κ. Μαγκίνε, η κυρία Μαγκίνε, με συγχωρείτε, ευχαριστώ δίνοντας συνέχεια σε αυτό το οποίο είπε ο σα, νομίζω ότι το θέμα της ισότητας, της δικαιοσύνης μεταξύ παραγωγών, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ανταγωνιστών είναι πολύ σημαντικό. Και ο τομέας των εγωπροβάτων έχει δυσκολίες όσοι είναι, οι κτηνοτρόφοι λένε στην Ιρλανδία ότι με την ηλεκτρονική καταγραφή ε, θα χρεοκοπήσουν και θα πρέπει να εγκαταλείψουν τα ζώα. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, να δούμε τι κάνουμε. Και επίση ε, έγιναν ορισμένε παραχωρήσεις, το παραδέχομαι, αλλά όσον αφορά την ισοτιμία. Είχαμε αυτό με το κρέσο από τη Βραζιλία και τώρα με την σήμανση ε, των εγωπροβάτων, αλλά όχι με τα ζώα από τρίτε χώρε. Επίση, πώς μπορεί ε, να, τα κράτη να βοηθήσουν στη σήμανση. Προτείνω λοιπόν ε, ενώ η Επιτροπή μας δεν μπορεί να σταματήσει αυτές τις εξελίξεις, θα μπορούσαμε τουλάχιστον να γράψουμε στο νέο πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας και της Επιτροπής Περιβάλλοντος και να του ζητήσουμε να λάβουν υπόψη τις ανησυχίες μας. Και εκείνοι θα μπορούσαν να το δουν αυτό το θέμα από διαφορετική σκοπιά. Αλλά οι αναφέροντες είχαν έλθει σε αυτή την Επιτροπή στο παρελθόν και αντιπροσωπεύουν πολλούς ανθρώπους ε, ε, στις χώρες όπου υπάρχουν πολλά εγώ πρόβατα, αλλά νομίζω ότι αυτή η τάση δεν θα σταματήσει. Ευχαριστώ κύριο Άτκινς. κυρία Άτκιν, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Ε, να ε, απαντήσω στα λόγια της κυρίας Μακίνες για Όσες βρισκόμαστε στο Λασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα, αργά το βράδυ με την κυρία Βασιλείου, μας είπε ακριβώς ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά τις εισαγωγέ από ε, τρίτες χώρες. Παραθέτω λοιπόν αυτά που είπε. Είπε ότι το μόνο που μπορούμε να απαιτήσουμε ε, είναι μέτρα τα οποία έχουν ισοδύναμες επιπτώσεις τα δικά μας. Και επίσης όσον αφορά την ειχνή συλλασιμότητα, ότι ο στόχος των κανόνων αυτών ε, είναι ε, πολύ, το εύρος είναι πολύ πιο περιορισμένο από ότι ο δικός μας. Και αυτό το ξεκαθάρισε και η Επίτροπος. Τέλος πάντων, για να επανέλθω τώρα στην την αναφορά, την οποία ε, την υποστηρίζω. Στην απάντηση της Επιτροπής αναφέρεται μία μελέτη που παρουσιάστηκε στη μόνιμη επιτροπή Και, τα λοιπά, και που είναι διαθέσιμη στην ε, ιστοσελίδα. Εγώ τη έριξα μια ματιά. Γιατί αυτή η μελέτη εξετάζει το κόστος Και νομίζω ότι όταν εξετάσει κανείς το κόστος θα καταλάβει ότι υπάρχει πλήρης έλλειψη αναλογίας με το αποτέλεσμα. Παράδειγμα, ε, στην ε, ε, σύνοψη αναφέρει ότι πάνω από 90% του κόστους, του σχετικού κόστους, θα τελικά πέσει στους ώμους των επιμέρους γεωργών. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι το κόστος είναι διαφορετικό ανάλογα με το κράτος μέλος. Και αυτό εξηγείται από διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, από το πόσα, πόσες είναι οι μικρές εκμεταλλεύσεις, το κόστος ε, του εξοπλισμού. Με δύο λόγια υπάρχει μεγάλη διαφορά ε, από τους κόστους όσον αφορά τα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω αν εδώ επισέρχεται κάποιο ζήτημα ιστορικής αγοράς, πάντως σίγουρα ενδιαφέρει ιδιαίτερα του επιμέρους ε, ε, γεωργούς σε μέρους κράτη-μέλη. Επίσης, το κόστος τη ηλεκτρονική αναγνώριση είναι 1,4 1,6 φορέ περισσότερο από ό,τι το συμβατικό σύστημα. Ποιο το πληρώσει αυτό το παραπάνω κόστο. Και τέλο, τελευταίο σχόλιο όσον αφορά αυτή την ενδιαφέρουσα αναφορά που όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το ζήτημα πρέπει να διαβάσουν και την ενδιαφέρουσα έκθεση. Αν εξετάσει κανεί το κόστο ε, εξοπλισμού και το κόστο ανάγνωση ε, και το εξετάσει από τη σκοπιά των εκμεταλλεύσεων, των σφαγείων και των δημοσίων υπηρεσιών, όσον αφορά το κόστο εξοπλισμού, Όσον αφορά τι επιμέρου εκμεταλλεύσει ε, και του επιμέρου γεωργού, εδώ τα πράγματα είναι ιδιαίτερα τα πανηρά, αλλά, ε, και δεν υπάρχει κανένα αντιστάθμισμα όσον αφορά ε, τα ωφέλη. Τα ωφέλη όλα τα εισπράττει η αγορά, οι δημόσιε υπηρεσίε κτλ. Άρα εδώ έχουμε πλήρη διατάραξη τη οροπία. Υποστηρίζω του αναφέροντε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί η εφαρμογή όλων αυτών, όπω πρότεινε ο κύριο Σμιθ. Εξαιρετική αυτή η ιδέα και υποστηρίζω και την άποψη της κυρίας Μαγκίνες να αποστείλουμε επιστολή ε, των Προέδρων ε, των Επιτροπών Γεωργίας και Περιβάλλοντος για να τονίσουμε τις απόψεις τους σε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Και κάτι άλλο. Επειδή σε όλους, σε όλους μας αρέσει να μιλάμε για τα δικά μας κράτη-μέλη, να δούμε τι γίνεται στην Ιρλανδία. Ο αριθμός των ζώων όλο και μειώνεται ε, και ένα τέτοιο μέτρο θα οδηγήσει σε θάνατο του κλάδου. Γιατί όσο πιο μικρό είναι το, όσο πιο μικρή είναι η εκμετάλλευση και το κοπάδι, τότε το το κόστο είναι μεγαλύτερο. Άρα τουλάχιστον στην Ιρλανδία αυτό θα σημάνει ότι θα καταστραφούν οι μικρέ εκμεταλλεύσει. Κύριε Ντεμπρότ. Και εγώ θέλω να συμφωνήσω με τους προηγούμενους συναδέλφους. Είναι σαφές από τον αριθμό συναδέλφων βουλευτών που έλαβαν το λόγο σήμερα εδώ και από αυτά που είπαν οι αναφέροντες και από το ότι πολλά κράτη-μέλη θίγουν αυτό το θέμα στο Συμβούλιο. Από όλα αυτά είναι σαφές ότι το θέμα αυτό πρέπει να επανεξεταστεί. Όπως είπαν οι συνάδελφοι, είμαστε ρεαλιστές. Ξέρουμε ότι η ημερομηνία πλησιάζει και ότι κάτι πρέπει να γίνει. Αλλά επειδή ακριβώς είναι τόσο σημαντικό το θέμα και απασχολεί τόσο πολύ κόσμο, κάτι πρέπει να γίνει με την επανεξέτασή του. Και όπως φαίνεται από την αναφορά αυτή και από τους ευρωβουλευτές που έλαβαν τον λόγο, φαίνεται ότι μας ενδιαφέρει το θέμα και θέλουμε να δώσουμε σημασία στα αιτήματα των πολιτών είναι ένα θέμα που πρέπει οπωσδήποτε να επανεξεταστεί. Κύριε Ζιά, ε, όπως ε, και οι προηγούμενοι ομιλητέ, ε, το ίδιο θέλω να πω και εγώ. Λέω το λόγο απλώς για να πω ότι και στη Γερμανία έχουμε τα ίδια προβλήματα. Έχουμε τομέα προβίου κρέατο και να γίνει η διάκριση μεταξύ των μικρών και των μεγάλων ε, προβάτων και ε, προσωπικά αν θέλετε με ενδιαφέρει ε, το θέμα αυτού του κλάδου. Έχουμε αρχίσει να συζητάμε αυτό το θέμα πριν από χρόνια και τώρα που πλησιάζει στο τέλος του το θέμα φαίνεται ότι αλλάζουν ε, οι θέσεις ε, και φαίνεται ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες ε, διατάξεις. Εμείς αναφέρουμε προς την Επιτροπή τα θέματα αυτά εφόσον έχουμε λάβει τις αναφορές των πολιτών. Αλλά νομίζω ότι είναι ανεπαρκής αυτή η διαδικασία και δεν αφορά μόνο το εγωπρόβιο κρέας. Νομίζω ότι ε, το κόστος θα είναι τεράστιο για όλο τον τομέα. και δεν ε, βλέπω να δικαιολογείται το κόστος έναντι των πιθανών ε, ωφελών. Άλλη μια φορά λοιπόν να ζητήσουμε από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ασχοληθούν με το θέμα αυτό. και προς εσάς θα ήθελα να ρωτήσω, Πρόεδρε, αν υπάρχει κάποια διατύπωση να ζητήσουμε από την Επιτροπή να εξετάσει αυτή την αναφορά υπό την έννοια του αιτήματο του αναφέροντος. Νομίζω ότι ε, στο τέλος αυτής ε, της συζήτησης, όπου τόσοι πήραν το λόγο για αυτή την αναφορά, μπορούμε πραγματικά να πούμε ότι δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Εκτός και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάτι να προσθέσει. Νομίζω ότι θα ήταν δυνατόν να προτείνουμε να ε, μεταφέρουμε την, να κοινοποιήσουμε την αναφορά στην Επιτροπή Γεωργίας για να τοποθετηθεί και η Επιτροπή αυτή και να δούμε μήπως θα μπορούσαμε να αναλάβουμε μία πρωτοβουλία. Γιατί νομίζω ότι η αρμόδια Επιτροπή είναι η Επιτροπή Γεωργίας. Αν λοιπόν δεν ε, διαφωνείτε, θα πρότεινα να ε, στείλουμε τα πρακτικά στην Επιτροπή Γεωργίας για να γνωμοδοτήσει. Σας ευχαριστώ και νομίζω ότι τώρα μπορούμε να περάσουμε στην 11 την ε, αναφορά ε, υπαριθμών 11-997 2007. Έχουμε δύο αναφέροντες, γιατί έχουμε δύο αναφορές και 15-18-2008. Είναι παρόντες. So the, screen on because he's going to, make a PowerPoint uh, presentation. Είναι παρόντες και οι δύο, και αναφέρον και αναφέρουσα. Ο Ιβαήλο Ιβάνοφ και η Ειρήνα Ματιέβα. Για να δούμε, ε, ζητούν, προσπαθούμε λίγο να εγκαταστήσουμε ένα ιδιαίτερα ε, ε, δύσκολο τεχνολογικό ζήτημα για την αίθουσα. Γι' αυτό ε, προτείνω να κάνουμε πέντε λεπτά διάλειμμα μέχρι να λύσουμε αυτό το τόσο δύσκολο πρόβλημα. Ευχαριστώ. Bene, se possiamo rimetterci a posto perché siamo... Μήπως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Να δώσω το λόγο στην κυρία Ματέβα. Μάλιστα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομη. διότι ίσως ε, ή, πήρατε την ενημέρωση από την BirdLife International και έχετε διαβάσει το κείμενο των ε, δύο αυτών αναφορών. Ε, το πρώτο αφορά την επάρκεια των ειδικών ζωνών προστασία στα πλαίσια τη ε, οδηγία ε, για τα πτηνά. Εγώ θα ήθελα επίση την προσοχή σα στο εξή. Μετά από πολλέ προσπάθειε που καταβάλαμε, προσπάθειες και από μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέχρι στιγμής έχουν γίνει αποδεκτές από την κυβέρνηση 114 περιοχές πτηνών ενώ 26 δεν έχουν γίνει δεκτές. Ε, και ε, οι περιφέρειες των έξι ονών μειώθηκαν σημαντικά. Κοιτάξτε, ε, δεν υπάρχει λοιπόν ο επαρκής βαθμός προστασίας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα σε σχέση με αυτές τις ζώνες μειωμένης προστασίας. Ε, εδώ βλέπετε ε, ένα από τα είδη αυτά, ε, το οποίο αποτελεί αντικείμενο προστασίας, Αιγυπτιακό όρνεο. Εδώ λοιπόν βλέπετε πως οι περισσότερες αυτές τις περιοχές βρίσκονται εκτός της προστασίας του Natura 2000. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο επιμένουμε για αυτές τις έξι ζώνες που μειώθηκαν σημαντικά να ε, ε, γίνουν δεκτές στο σύνολό τους και να μην έχουμε αυτή τη μείωση. Αυτό είναι ένα από τα παράδειγμα μειωμένων περιοχών. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην Καλιάκρα. Και ε, αυτή η περιοχή συνδέεται με τη δεύτερη αναφορά. Βλέπετε εδώ την περιοχή που αποκλείεται, βλέπετε στη διαφάνεια. Εδώ η λευκή πελαργή και άλλα ε, πτηνά συγκεντρώνονται, οι χήνες ε, και ε, ε, ένα, ένα είδος χήνας που έχει κόκκινο στήθος και αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί σε αυτές τις περιοχές γίνονται αναπτυξιακές δραστηριότητες, τουριστικής φύσεως, αιωλικά πάρκα κτλ. Αν εφαρμοστούν τελικά και γίνουν όλα αυτά τα σχέδια, μεγάλο μέρος των ζωνών θα ε, εξαιρεθεί, θα καταστραφεί. Τώρα, ε, πάρκα, τι εννοώ. Τι γίνεται στην Καλλιάκρα. Τελικά θα καταστραφούν τα οικοσυστήματα κατά, την, δραστηρι... κατά τις δραστηριότητες αυτές. Επιπλέον, ένα από τα αιωλικά πάρκα που κατασκευάστηκε πριν από αρκετό καιρό. Τον πρώτο χρόνο που άρχισε να λειτουργεί είχαμε ε, θανατώσεις πτηνών. Βλέπετε εδώ τον πελεκάνο, συγκεκριμένα ένα είδος πελεκάνου και δυστυχώς δεν είναι το μόνο θύμο. Ενάμιση χρόνο αργότερα, ε, ενάμιση χρόνο δηλαδή μετά την κατασκευή των αιωλικών πάρκων, είχαμε αυτά τα τρομερά αποτελέσματα. Και αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι ε, αυτή, ε, ε, αυτή η τάση επαναλαμβάνεται παρά τους ευθυρότατους περιορισμούς. Στις περιοχές, ακόμα και στις περιοχές που δεν βρίσκονται στο Natura 2000, θεωρούμε ότι όπου κατασκευαστούν ολικά πάρκα θα δημιουργηθούν τα ίδια προβλήματα. Το βλέπετε εδώ στη διαφάνεια. Και χαιρόμαστε και εκτιμούμε ιδιαίτερα τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί έστειλαν ε, προειδοποιητικές επιστολές. Αλλά δεν αρκούν όλα αυτά. Επειδή συνεχίζονται αυτά τα καταστροφικά αποτελέσματα στην περιοχή, ε, η νεοεκλεγική ε, κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι θα υπάρξει απόλυτη διαφάνεια και θα υπάρξουν αυστηρότατα μέτρα. εναντίον ε, των ανθρώπων που διαπράττουν αντικείμενα και παραβιάζουν τον νόμο. το νόμο ε, εννοώντα και τη βουλγαρική νομοθεσία αλλά και την κοινωτική νομοθεσία, οδηγία για τα πτηνά και τα οικοσυστήματα. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι για μας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει ε, και η Επιτροπή μάλλον αναφορά θα πρέπει να ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, απευθύνει έκκληση τελικά προς τις αρχές της Βουλγαρίας. Ε, όχι προειδοποίηση, έκκληση να, να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα όσο να πιο γρήγορα για να σταματήσουν αυτές οι καταστροφές. και να υπάρξει πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Γιατί δεν έχουμε καμία εγγύηση για το ότι θα προστατεύονται πραγματικά αυτές οι περιοχές. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριος Παπούλιας. Παπούλια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ έχουμε την αναφορά υπαριθμών 997 και για τη δεύτερη αναφορά θα μιλήσει κάποιος άλλος συνάδελφός μου. Αυτή η αναφορά, αφορά το ότι δεν υπάρχει πλήρης εθνικός κατάλογος ε, ε, ε, τόπων Natura 2000 στη Βουλγαρία, είναι μια αναφορά που έγινε το 2007, και ευτυχώς πρέπει να πω ότι από το 2007 έχουν εξελιχθεί θετικά τα πράγματα και ήδη τώρα στη Βουλγαρία Υπάρχει ένας ε, κατάλογος ε, σημείων προστασίας ε, με βάση το δίκτυο Natura 2000. Βέβαια ανησυχεί ακόμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί υπάρχουν πολλά κενά στον κατάλογο της Βουλγαρίας και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να συνομιλεί με τις βουλγαρικές αρχές για να καλυφθούν αυτά τα κενά που υπάρχουν στον κατάλογο. Πιο συγκεκριμένα αφορά την οδηγία για τα ενδιατήματα. Οι αξιολογήσεις που έχουν γίνει για αυτές τις περιοχές κοινοτική σημασίας που συζητούνται με βάση αυτήν την οδηγία βασίζονται στην βιογεωγραφική ανάλυση που έχει δοθεί και στις βουλγαρικές αρχές και οι βουλγαρικές αρχές προετοιμάζουν την απάντησή τους προς την Επιτροπή προσπαθώντας να καλύψουν τα υπάρχοντα κενά. Πρέπει να πω ότι το 30% της επικράτειας της Βουλγαρίας καλύπτεται από τέτοιες περιοχές κοινοτικής σημασίας και δεν μένουν ακόμη πολύ σημαντικά κενά. Τα κενά όμως που υπάρχουν αναμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα αντιμετωπιστούν και περιμένουμε από τη Βουλγαρία την πλήρη απάντησή της για το θέμα αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά τοποθεσίε που θα πρέπει να χαρακτηριστούν ω ζώνε ειδική προστασία βάσει τη οδηγία για τα πτηνά, οι βουλγαρικέ αρχέ ήδη καλύπτουν ε, τον επιστημονικό κατάλογο με τις σημαντικές περιοχές, τον κατάλογο που προετοίμασε η BirdLife, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμη ανησυχεί διότι λείπουν κάποιες σημαντικές περιοχές από τις περιοχές που ορίστηκαν ε, ειδική προστασίας. Αυτές είναι οι περιοχές που αναφέρθηκαν και από τον αναφέροντα, έξι βασικές περιοχές. Και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το θέμα με βάση και μια διαδικασία παραβάση που ξεκίνησε κατά της Βουλγαρίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει και ζητάμε τα ε, πλέον επίκαιρα επιστημονικά δεδομένα για να αξιολογήσουμε την οικολογική σημασία αυτών των περιοχών. Αναμένουμε μέχρι τα τέλη του 2009 πλήρη απάντηση από τις βουλγαρικές αρχές και τότε θα αποφασίσουμε για τη συνέχιση που θα δοθεί σε αυτή τη διαδικασία παραβάση. Ακόμη αναφέρονται, αναφέρουν τα θέματα προστασίας των περιοχών και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα, καλυ... θα καλυφθεί από το συνάδελφο με βάση τη δεύτερη αναφορά για το ίδιο θέμα. Ευχαριστώ. Ε, thank, thank you, Mr. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Παπούλιας ανέφερε ότι έχει αρχίσει μια διαδικασία επιπαραβάση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της μη πληρότητας του δικτύου ζωνών ε, ειδική προστασία στη Βουλγαρία. Και όπως αναφέρει ήδη η αναφέρουσα, η Επιτροπή έχει ξεκινήσει και διαδικασία επιπαραβάση για κάποια θέματα ε, τοπικής ανάπτυξης ε, και κάποια προγράμματα ανάπτυξης σε αυτές τις περιοχές που αναφέρονται από την αναφέρουσα. Έχει αρχίσει μια διαδικασία επιπεραβάσης συγκεκριμένα για το Καλλιάκρα. την περιοχή για την οποία μας δόθηκαν και κάποιες εικόνες προηγουμένως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει την ανησυχία της για τη σωρευτική επίπτωση των αιωλικών πάρκων στις συγκεκριμένες αυτές περιοχές. Έγιναν κάποιες συζητήσεις και με τις βουλγαρικές αρχές και οι βουλγαρικές αρχές μας είπαν ότι εξετάζουν τώρα την ιδέα μιας ε, παύσης των περαιτέρω δράσεων ανάπτυξης σε αυτή την περιοχή στο, και ότι έχει ολοκληρωθεί μια στρατηγική μελέτη επιπτώσεων που έχει ως σκοπό να αντιμετωπίσει συνολικά το θέμα της ανάπτυξης αιωλικής ενέργειας και χαρακτηρισμού αυτών των περιοχών. Η Επιτροπή υποστηρίζει την ανάπτυξη αιωλικής ενέργειας στη Βουλγαρία αλλά θέλουμε η σχετική ανάπτυξη να γίνεται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η αντιπαράθεση με τους στόχους της οδηγίας για τα πτηνά. Η Επιτροπή σας μπορεί να είναι ησυχή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να αποδίδει την πρέπουσα σημασία σε αυτό το θέμα και θα σας ενημερώνουμε για τις περαιτέρω εξελίξεις σε σχέση με την διαδικασία επιπαραβάση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να λάβω το λόγο για να πω δύο λόγια για την νομική προστασία αυτών των περιοχών και για τα μέτρα που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά. Ε, καταρχήν, η νομική προστασία των περιοχών που δεν έχουν χαρακτηριστεί πλήρως ως ζώνες ειδικής προστασίας. Υπάρχουν τέτοιες περιοχές που θεωρείται ότι προστατεύονται και η προστασία χορηγείται βάσει της εθνικής νομοθεσίας. Όμως αυτές οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν τηρούνται και γι' αυτό ξεκινήσαμε μια διαδικασία παραβάση κατά της Βουλγαρίας για συστηματική παραβίαση του ε, καθεστώτος προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας για τα Πτηνά και θέλουμε να αποφύγουμε την επιδείνωση της κατάστασης της περιοχής και τις ενοχλήσεις προς τα πτηνά. Επίσης, έχουμε ξεκινήσει και άλλες διαδικασίες επί παραβάση και μπορούμε να πούμε ότι ε, υπάρχουν κάποιες ε, ανησυχητικές εστίες στη Βουλγαρία, στον εύξηνο πόντο και στις ορεινές περιοχές και καλύπτονται αυτές τις περιοχές από διαδικασίες επί παραβάση αυτή τη στιγμή. Και προς το παρόν, όπως είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, σε συζητήσεις με τη βουλγαρική κυβέρνηση και με μη κυβερνητικές οργανώσεις, είδαμε ότι προσπαθεί η κυβέρνηση τώρα να διασφαλίσει καθεστώς προστασίας για τις περιοχές αυτές και να συνεχίσει με την ολοκλήρωση του χαρακτηρισμού των περιοχών δικτύου Natura 2000 στη Βουλγαρία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο στον επόμενο μιλητή, στην κυρία Γιωτόβα. Тревожно е, че един такъв проблем, който е поставен още през 2007 година, все още... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αρχίσαμε να το συζητάμε το θέμα αυτό το 2007 και ακόμη δεν έχουμε κάποια τελική απάντηση. Ακούμε ότι όντω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταβάλει πολλές προσπάθειες για την επίλυση του θέματος, αλλά δεν έχουμε ακόμη απτά αποτελέσματα δεν μιλάμε μόνο για περιοχές ειδική προστασίας και για διατήρηση της πανίδας και χλωρίδας. Μιλάμε για τη διατήρηση ειδών τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση. Μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες ακροάσεων, διαδικασία επιπαραβάση κλπ θα χαθούν όλα αυτά τα είδη τα οποία σας λέω ότι διατρέχουν τον κίνδυνο εξαφάνισης. Είδαμε κάποιες εικόνες και σας διαβεβαιώ ότι υπάρχουν και εικόνες που είναι ακόμη πιο τρομακτικές και ανησυχητικές από αυτές που είδαμε. Προτείνω να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη γνώμη έχει. Μέχρι τώρα από την βουλγαρική κυβέρνηση είχαμε απλώς υποσχέσεις. Δεν ξέρουμε τι έχει όντως εκπληρώσει από όλες αυτές τις υποσχέσεις. Και θα περιμένουμε και σχετικές πληροφορίες στην αρχή του επομένου έτους. Γιατί η προθεσμία για την υποβολή πληροφοριών από τη βουλγαρική κυβέρνηση τελειώνει στα τέλη του 2009 και μετά μπορούμε στην Επιτροπή να αποφασίσουμε τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα για να παρέμβουμε. Όντω, περίπου το 30% της, της επικράτειας της Βουλγαρίας προστατεύεται από το Natura 2000, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τις αμελεί αυτές τις περιοχές η βουλγαρική κυβέρνηση. Και υπάρχει και άλλο ένα σημείο που θεωρώ σημαντικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθούν τη σωστή εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να επιβληθεί πιο αυστηρή παρακολούθηση στη Βουλγαρία γιατί δεν μιλάμε μόνο για παραβίαση εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, μιλάμε για κάτι ακόμη πιο σημαντικό. έχουμε διατάξεις που δεν τηρούνται από τις τοπικές ή εθνικές αρχές και υπάρχουν και τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών, πολυεθνικών εταιριών και εταιριών που ασχολούνται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λέμε ότι είναι σημαντικές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, αλλά δεν θα πρέπει να παραβιάζεται η νομοθεσία. Κάνω έκκληση λοιπόν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σας παρακαλώ να ασκήσετε ακόμη πιο αυστηρό έλεγχο για τις δραστηριότητες της βουλγαρικής κυβέρνησης. Ευχαριστώ. κυρία Ντεμπρούν. Ευχαριστώ πολύ. Έκανα ένα γραπτό ερώτημα στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών ερωτήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα της μη της μη προς την οδηγία για τα πτηνά και ιδίως για το χαρακτηρισμό ζωνών ειδικής προστασίας. Αφού έχω κάνει λοιπόν την ερώτησή μου, το αφήνω στην Επιτροπή, αφού το έχω ήδη ζητήσει. Και σήμερα θέλω συγκεκριμένα να μιλήσω όχι τόσο για το χαρακτηρισμό ζωνών, αλλά για την υλοποίηση των μέτρων. Θέλουμε να λάβει μέτρα η Επιτροπή και να το παρακολουθεί το θέμα με τις βουλγαρικές αρχές γιατί ο κίνδυνος συνεχίζει να υπάρχει και χάνουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή αν μπορεί να επιταχύνει τις διαδικασίες την παραβάση. Όταν οι βουλγαρικές αρχές λένε ότι σκέφτονται το ενδεχόμενο παύσης αυτών των δραστηριοτήτων, ε, τι εννοούν, πότε θα το σκεφτούν και πότε θα εφαρμόσουν ένα μορατόριο ε, για, αυτά τα προγράμματα τα αναπτυξιακά. Υπάρχει δυνατότητα να σταματήσουν αυτά τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται παρότι υπάρχει διαδικασία παραβάση για να αποφύγουμε την καταστροφή την οποία μας περιέγραψαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Ευχαριστώ. Merci, Madame la Présidente. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. σύμφωνα με τους προηγούμενους συναδέλφους, θα ήθελα και εγώ να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά, χωρίς να επαναλάβω τα όσα υπόθηκαν ήδη. Απλά και μόνο θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό το σημείο ότι το βουλγαρικό κράτος πρέπει να επιδείξει καλή θέληση. Είναι μεν κάτι, αλλά δεν αρκεί το να πούμε το 30% της βουλευτικής επικράτειας είναι ανοιχτή, ε, αυτό δεν είναι επιχείρημα και όχι επιστημονικό επιχείρημα. Και όχι, επιχείρημα που καταδεικνύει ότι οι στόχοι της οδηγίας οικοτόπων ή πτηνών που πρέπει να έχει αντικείμενο να εξασφαλίσει την καλή διαφύλαξη των ειδών που αναφέρονται στις οδηγίες. Αυτό το επιχείρημα όμως σήμερα δεν μπορεί να μας πείσει και να μας διαβεβαιώσει ότι το βελγικό κράτος συμμετέχει στη στρατηγική για την καταπολέμηση της απόλυσης βιοπικιλότητας και ότι σήμερα βρίσκεται στο ύψος των στόχων αυτών. Επίσης συμφωνώ με τον προβληματισμό. Όταν μας λένε ότι η Βουλγαρία δεν σέβει τις υποχρεώσεις της, ότι οι διαδικασίες παραβίασης έχουν ξεκινήσει, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα πράγματα για να εμποδίσουμε ή να επιβραδύνουμε την καταστροφή των δύο τόπων και των προστατευμένων ειδών. Αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι έχουμε να κάνουμε με ένα αγώνα ταχύτητος. Τι θα συμβεί, τι μπορούμε να κάνουμε ακόμα όταν οι ιδιότοποι και κυρίως αυτοί οι χώροι που βρίσκονται στη Μαύρη Θάλασσα κοντά θα ε, χτιστούν. Τι θα πούμε, ε, θα διαπιστώσουμε την παραβίαση, θα επιβάλλουμε κυρώσει, τι θα κάνουμε. Τελικά οι στόχοι ε, της οδηγίας ε, των βιοτόπων και των πτηνών δεν θα έχουν γίνει σεβαστοί. Συμφωνώ λοιπόν με τι παρατηρήσεις που έγιναν. Τι μπορούμε να κάνουμε, έστω ε, συμβολικά ή πολιτικά για να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα στο, βελγικό ε, στο βουλγαρικό κράτος, να τους επαναφέρουμε στη λογική ώστε να αρχίσουν να εφαρμόζουν την οδηγία των βιοτόπων και πτηνών. Ευχαριστώ κύριε Μπουσινάρου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Aceste petiții sunt uh, valabile nu doar în cazul Bulgariei. Λοιπόν, όσον αφορά τι μεταφορέ αυτέ, αυτέ δεν αφορούν μόνο τη Βουλγαρία, μην το ξεχνάμε. Τέλο πάντων, ξαναγυρίζω στο θέμα των δύο αυτών αναφορών. Νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον δύο πράγματα. Να πάρουμε επικαιροποιημένε πληροφορίε πληροφορίες για την κατάσταση στη Βουλγαρία όσον αφορά τις ε, ε ειδικέ ζώνες προστασίας. Πληροφορίες λοιπόν και ενημέρωση από την κυβέρνηση Βουλγαρίας και ενημέρωση από την Επιτροπή. Γιατί οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής παραπέμπουν ε, στην κατάσταση του 2008. Και μέχρι να πάρουμε όλε αυτέ τι πληροφορίε, να κρατήσουμε ανοιχτέ τι αναφορέ. Και τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έχουμε και μία έκθεση ιδία πρωτοβουλία για την βιοπικιλότητα στην Επιτροπή μας. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να διατυπώσουμε ένα σύνολο κανόνων όσον αφορά τις συνθήκες για την εγκατάσταση ολικών πάρκων. Η έλλειψη πληροφορίας και νομοθεσίας στο συγκεκριμένο τομέα δημιουργεί τρομερά προβλήματα. Πίσω από αυτά τα ολικά πάρκα βρίσκονται εταιρείε όπως η ΕΟΝ στη Γερμανία, οι ηλεκτρισιτές στην Γαλλία και ε, ε, πραγματικά είναι πολύ περιορισμένε οι δυνατότητες της τοπικής αυτοδιοίκηση αλλά και των κεντρικών κυβερνήσεων. Εκτός και αν υπάρχει νομοθεσία που να ισχύει για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και να υπάρξουν και ε, δεσμευτικές ε, ημερομηνίες και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο θα πρέπει να τηρηθεί από όλου, Μιλώ για, τις, για την περιβαλλοντική αξιολόγηση αν δεν ε, υπάρξει λύση προ την κατεύθυνση αυτή, θα αντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα. Τα ίδια προβλήματα έχουμε και εμεί στη Ρουμανία με τα αεολικά πάρκα. Και σε μία κρόαση που έγινε πρόσφατα ε, στην ε, Επιτροπή Ρέτζι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα είπε ότι μέχρι στιγμή υπάρχουν παραθυράκια στην νομοθεσία. Πρέπει λοιπόν να, να ρυθμίσουμε τα πράγματα, να λύσουμε την κατάσταση και εμεί, η Επιτροπή Αναφορών, είμαστε αρμόδιοι για, ε, τη, και θα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες υποδείξεις για να βοηθήσουμε την Επιτροπή να διατυπώσει αυτό το σύνολο κανόνων. Σύντομα θα έχουμε τη νέα Επιτροπή με ατζέντα η οποία ε, θα είναι τελική στους επόμενους 6 μήνες. Αλλά στο μεταξύ θα τα, ε, τα ίδια αυτά ε, απειλούνται με αφανισμό. Ευχαριστώ. Okay. Oh, ε, Αν μου επιτρέπετε. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Και με το φόβο να μην εστιάζομαι ε, στα σχέδια κατασκευής ελικών πάρκων. Εάν ε, χρειάζεται να έχουμε συγκεκριμένους κανόνες, κυρίως ε, τον κανονισμό που καταστρέφει το κεφάλαιό μας της βιοποικιλότητας, αυτό ισχύει με τον ίδιο τρόπο. Δεν πρέπει να εστιάζουμε στα αιωλικά στην ολική ενέργεια. Αυτό αγγίζει όλες τις ακτές της Ευρώπης. Υπάρχουν ορισμένα διαμάντια, ε, φυσικά διαμάντια, τα οποία αυτή τη στιγμή υπονομεύονται από πολεοδομικά σχέδια και νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικό πρόβλημα και πρέπει να δούμε πώς, κατά πόσο είμαστε ικανοί να αξιοποιούμε αυτό το φυσικό κεφάλαιο που υπάρχει κυρίως ανατολικά της Ευρώπης στις νέες χώρες που προσχώρησαν και αυτή τη στιγμή καταστρέφεται, υπονομεύεται πλήρω. Øh, øh- Αν μου επιτρέπετε να πω το εξή. Τα περισσότερα από τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνοι. Νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτέ αυτέ τι αναφορέ. Αλλά να προσθέσουμε και κάτι άλλο. Κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό της Βουλγαρίας, για τη Βουλγαρία είναι το γεγονό ότι οι πολίτε είναι ιδιαίτερα δραστήριοι, λαμβάνουν, παίρνουν την κατάσταση στα χέρια του. Ε, αναλαμβάνουν συγκεκριμένη δράση. Και αυτό ε, μα συμφέρει όλου. Πραγματικά ε, είναι προ όφελο όλων μα το γεγονό ότι είναι τόσο δραστήριοι οι πολίτε τη Βουλγαρία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και να πω και κάτι άλλο. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να συνδέουμε το ζήτημα μόνο με τα αιωλικά πάρκα. Ε, και βεβαίως το ζήτημα αυτό το συζητάμε ε, στη, ε, στη χώρα μας. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα μπορούν να έχουν αντίκτυπο επιζήμιο για το περιβάλλον. Οι παραφεριστικές κατοικίες, για παράδειγμα και σε πολύ πιο μόνιμη βάση. Έχουμε λοιπόν το ζήτημα αυτό το οποίο προκύπτει με τι ανανεώσιμε ενέργειε. Και βεβαίω πρέπει να είμαστε πολύ προκτικοί Ε, αλλά ε, καταλαβαίνω ότι τα προβλήματα αυτά ε, που με τα φτηνά είναι πρόβλημα και για τη χώρα μας. Δηλαδή, όταν όμως τα, τα πτηνά ε, συνηθίσουν τη νέα πραγματικότητα, τότε πραγματικά τα πράγματα αλλάζουν. Ναι, μην μη συγκρίνουμε όμως τα ολικά πάρκα ε, με την ε, ε, μαζική κατασκευή κατοικιών. Γιατί στην πρώτη περίπτωση μπορούμε να αφαιρέσουμε τις ανεμογεννήτριες, στη δεύτερη περίπτωση οι κατοικίες είναι μόνιμες. Δεν υπάρχει δρόμος, του, δεν υπάρχει δρόμος προς τα πίσω. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κερδοσκοπικές τάσεις και τις δύο περιπτώσεις. Αν όμως είναι σωστός ο σχεδιασμός αυτής εξ αρχής, τότε δεν είναι και το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί για το περιβάλλον οι καινούργιες ανεμογεννήτριες ε, προκαλούν πολύ λιγότερες ε, ζημιές. Ε, είναι πολύ πιο... κάνουν πολύ λιγότερο θόρυβο από τις παλιές, είναι διακριτικότερη η παρουσία τους. Και σας το ξαναλέω, μπορούμε να τις αφαιρέσουμε και δεν αφήνουν μόνιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο διατηρούμε την αναφορά ανοιχτή. Νομίζω ότι αυτό ήταν η βούληση όλων των συναδέλφων που πήραν το λόγο. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε στον κύριο Μπουσινάρου ότι ίσως θα μπορούσε ε, να εκφράσει δικές του σκέψεις σε αυτή τη γνωμοδότηση στην οποία αναφέρθηκε. Και με αυτόν τον τρόπο θα την εμπλουτίσουμε. Δηλαδή, ε, με τη γνωμοδότησή μας να μεταφέρουμε αυτές τις απόψεις που ήδη έχει ξεκινήσει ε, η επεξεργασία και να κάνουμε και τις ε, περαιτέρω υποδείξεις στην αρμόδια επιτροπή. Όσον αφορά τώρα τις πιο κατάφορες παραβιάσεις που θα πρέπει να ξεκινήσουμε δικαστική δράση για να παρεμποδίσουμε αυτές τις ενέργειες, ίσως θα μπορούσε να υπάρξει και προσφυγή ενώπιον του δικαστηρίου για να σταματήσουμε αυτές τις δραστηριότητες πριν πολύ αργά. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να εργαστούμε με βάση την υπόθεση αυτή και αν συμφωνείτε όλοι να κλείσουμε το θέμα. Ε, non c'è nessun altro, va bene? Perfetto. Allora. Δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Ωραία. Al punto successivo και πάμε στο 12. Punto 12 sono iscritti. Στο 12 έχουμε διάφορες αναφορές. 683-2005 Βιντσέντσο Μαρμόρα. 31-2006 Τζαμπιέρο Άντζελη. 26.007 Μόνικα Σέπε 756.007 Τζοβάνι 789.007 789-2007 Τζίλιο Λαΐτσο 910-2007 Φραντσέσκο Ντι Πασκουάλε 991-2007 Βιντσέντσο Γκάλα 12-2008 Φραντσέσκο Μιλίνο από ένα πολίτη που δεν θέλει να αναφέρει το όνομά του στην ημερήσια διάταξη. 209-2008 Σεμπαστιώνα Περόνε. 347-2007 Τομάζο Εσπόστο και Βιρτζίνια Πετρελέζε. 587-2007 Μαρίνα Σαλβαντόρε. 1082-2008 Ραφαέλα Πατσίλιο. 396-2009 φατωνε Φατόνε. 12-23-2009 Ντανιέλε Τζόβε. Και θα προσέθετα και την, το θέμα 13, 955 2008 και 1011-2008 που αφορούν και αυτές οι δύο τελευταίες ε, αναφορές ε, τη διάθεση αποβλήτων ε, στην Ιταλία. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον πρώτο από τους υπογράφοντες που είναι παρόν, στην κυρία Μόνικα Σέπε. Grazie, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πραγματικά αισθάνομαι μεγάλη τιμή ε, που προσκλήθηκα στην Επιτροπή σας και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να συμμετάσχω. Το θέμα των αποβλήτων στην Καμπανία και ιδιαίτερα η απόφαση της κατασκευής ε, ε, ε ενός χώρου υγειονομικής ταφής ε, στη Βάλε Λαμασέρια, στην, στο Σαλέρνο, πραγματικά έχει πάρει μια πολύ δυσάρεστη τροπή. Πρέπει να πω ότι η λέξη επίγουσα ανάγκη σημαίνει το ίδιο σε όλες τις γλώσσες. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν γιατί στην καμπάνια παίρνει ένα διαφορετικό νόημα. Ε, η κυβέρνηση και η έκτακτη επιτροπή ε, πραγματικά έχουν ε, χρησιμοποιήσει τον όρο αυτό για να δικαιολογήσουν τις επιλογές τους. Φαίνεται λοιπόν ότι παρά τα νομοθετικά διατάγματα τα πάντα επιτρέπονται. Ε, ε, το, από το 2007 όμως ε, βρίσκονται απέναντι σε μια κοινότητα ανθρώπων που πραγματικά δεν θέλει αυτές τις προοπτικές ανάπτυξης που προέρχονται από αυτές τις δράσεις. θέλει να σεβόμαστε τους νόμους στην Ιταλική επικράτεια. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το σχέδιο του υγειονομικής σταφής στη Βάλε Ντελαμασέρια πραγματικά έχει δημιουργήσει τρομερά προβλήματα πώς πραγματικά ε, δεν, μπορούμε, ε, δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη οι στοιχειώδεις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος. Ε, μιλάμε για ένα υγρότοπο ο οποίος έχει διεθνή σημασία. Ε, που δίνει ζωή ε, σε ένα, ε, σε ένα σημαντικό οικοσύστημα, όπου, έχουν, όπου είναι παρόντα είδη, κοινοτικού ενδιαφέροντος, σε μια περιοχή που είναι καταφύγιο άγριων ζώων στα πλαίσια WWF, στο Περσάνο κτλ. Όλα αυτά δεν απέτρεψαν την κυβέρνηση της Ιταλίας από το να δημιουργήσει αυτό το χώρο υγειονομικής ταφής. Στο μεταξύ, σε περίπου 3 χιλιόμετρα απόσταση, πιο συγκεκριμένα, στο δάσος του Μάκια Σοπράνα, ε, το οποίο έχει έκταση περίπου 100 εκταρίων, ε, προφανώς, με ένδειξη του τότε Υπουργού Περιβάλλοντος, Πεκοράρο Σκάνιο, ε, θεωρούσαν ότι ε, το να, πραγματικά το να, ε, το, να αποψηλώσει το δάσος κατά 6 εκτάρια δεν σημαίνει και τίποτα. Και μιλάμε για ένα δάσος το οποίο ήταν σε μια εξαιρετική κατάσταση και που αποψηλώθηκε για πάντα. Δεν στάθηκαν ούτε για ένα δευτερόλεπτο να σκεφτούν πόσο παράλογη ήταν η απόφαση αυτή. το, το, πιο, το, το πιο σημαντικό ήταν η πόλη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας να απαλλαγεί από τα απόβλητα. Μέχρι στιγμή ε, μιλάμε για 700.000 τόνου ε, και άλλα τόσα θα έχουμε μέχρι τον Ιανουάριο 2010. Ε, πρόκειται για μια καταστροφή η οποία ήδη έχει ανακοινωθεί εδώ και καιρό και που ε, σημαίνει, ε, η, σημαίνει ε, μεγάλη, μεγάλη κερδοφορία για, για ορισμένους. μιλάμε για τη μαφία της δημόσιας διοίκησης και για ορισμένους νόμιμους εντός εισαγωγικών επιχειρηματίες. Ε, μιλάμε για το χάος, ε, για ε, πλήρη έλλειψη νομιμότητας στο Νότο και όλα αυτά δεν είναι τυχαία, αλλά μιλάμε για το αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο αναπτύχθηκε ο καπιταλισμός στην Ιταλία. Εδώ και δύο χρόνια πραγματικά υφίσταται τρομερά δεινά οι κάτοικοι της περιοχής. Δεν μπορεί μια κοινότητα 4.000 ε, κατοίκων να υφίσταται την έλλειψη πολιτισμού μιας ε, Μητρόπολης. Ε, σε αυτή, την, ε, σε αυτή την, την παράλογη ιστορία, εγώ δεν αισθάνομαι Ιταλίδα πολίτης, αλλά Ευρωπαία πολίτης. Ακριβώς γι' αυτό ήρθα εδώ, για να υπερασπιστώ και να υποστηρίξω το δικαίωμα στην αξιοπρέπειά μου. εάν δεν τιμωρηθεί η Ιταλία, σημαίνει ότι αύριο τα απόβλητα θα, μπορέσουν, θα, θα μπορούν πλέον να διατίθενται στο Κολοσσέο. Όμως ε, αυτό ε, μπορεί να είναι και πιο εύκολο με την έννοια ότι το Κολοσσέο τελικά δεν δίνει οξυγόνο ε, στους φτωχού πολίτες της χώρας μας. ευχαριστώ για την ε, υπομονή σα. Grazie. Σας ευχαριστώ. Successivo firmatario presente è la signora Gioiola Izzo. Buonasera.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 Καλημέρα. Σας ευχαριστώ σε όλους, ευχαριστώ τους φίλους της Επιτροπής ε, ε, που μου επέτρεψαν να εκφράσω ε, την θέση μου. Για μένα πρέπει να σας πω ότι αποτελεί ε, ιδιαίτερο ε, λόγο ικανοποίηση. Το γεγονό ότι βρίσκομαι εδώ σήμερα. Για εσά αυτό αποτελεί μια φυσιολογική άσκηση δημοκρατική συμμετοχή. Για μένα όμω είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονό, διότι ακριβώ ε, δείχνει το πόσο σημαντική είναι η δημοκρατία σε αντίθεση με αυτά τα οποία ε, ζούμε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μου. Λυπάμαι που μιλώ κατά τη χώρα μου, αλλά σα μιλώ για καταστάσει που έχουμε ζήσει όλοι. Δύο χρόνια έχουν περάσει από τότε που ε, έγιναν τα γεγονότα αυτά τα οποία καταγγέλλω και στην, και στην αναφορά μου και ζητώ την απονομή δικαιοσύνη, έτσι ώστε να προκύψει η αλήθεια για την περιοχή μα, η αλήθεια όσον αφορά την κατάσταση τη υγεία μα αλήθεια η οποία αποσιωπάται λόγω ε, αδράνειας ή λόγω, ε, ή ανεπάρκειας που ε, χαρακτηρίζεται από την κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την έλλειψη ευθύνης αυτών που υποτίθεται ότι προστατεύουν τα δικαιώματά μας. και τελικά ε, όλοι αυτοί που θα έπρεπε να είναι στο πλευρό μας για να καταπολεμήσουμε αυτούς που κυριαρχούν επί τόπου ε, και που καταπατούν τόσο κατάφορα τις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος με τα τοξικά αυτά απόβλητα. Επιτρέψτε μου να σας πω δύο λόγια για να καταλάβετε τι ακριβώς αποτελεί τη βάση της καταγγελίας μου. Γι' αυτό να σας ε, δώσω μια εικόνα ε, για την πραγματικότητα. Και βεβαίως θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο. Ζω σε μια μικρή πόλη 30.000 κατοίκων ε, στο νότιο-ανατολικό τμήμα τη Νάπολη, η οποία γειτονεύει με την Ατσέρα και με την Όλα. Ε, με τι οποίε περιοχέ τα τελευταία χρόνια ε, μοιραζόμαστε αυτή την κοινή, το γεγονό ότι βρισκόμαστε στο τρίγωνο του θανάτου. Σα σας παραπέμπω στο Lancet Oncology, στον τόμο 5, Τεύχος 9 του Σεπτέμβριου 2004, όπου αναφερόταν το τι ακριβώς συμβαίνει επί τόπου και ε, αποδεικνυόταν η κατάσταση περιβατολογικής ρήπανσης. Είναι πάρα πολύ σοβαρή. Σας παραπέμπω σε ορισμένα έργα κινηματογραφικά, τα οποία προσπαθούν να δείξουν τι ακριβώς γίνεται. Σας παραπέμπω στο έργο Gomorrah ή στο Beautiful Country, που μιλούν ακριβώς για αυτές τις παράνομες απορρίψεις αποβλήτων. Το Μαριλιάνο, η πόλη μου, κάποτε χαρακτηριζόταν από μια ανθίζουσα γεωργία, όπω άλλωστε και οι γειτονικέ χώρε. Ήταν ιδιαίτερα έφορη η γη μα και γι' αυτό ε, πραγματικά είχαμε τον τίτλο του Καμπάνια Φέλιξε, τη ευτυχισμένη γη. Μετά από μια κρίση της γεωργίας, η γη μας εγκαταλείφθηκε και τελικά κατάντησε να είναι χώρος ε, παράνομης διάθεσης ε, διαφόρων αποβλήτων. Και ε, όλα αυτά βεβαίως εμποδίζουν τη χρήση της γης και την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Ο προσωρινός χώρος αποθήκευσης ε, που επέβαλε με τη βία σε αρχές 2008 η έκτακτη επιτροπή της ε, κυβέρνησης δεν έλυσε το πρόβλημα, απλά και μόνο επιδίνωσε μια περιβαλλοντική κατάσταση που ήταν ήδη πολύ σοβαρή. Ε, τότε, το Φεβρουάριο του 2008, ήρθε στο φως μια υπόγεια δεξαμενή στα 30 μέτρα βάθος ε, και μάλιστα αυτό φάνηκε και μέσα από κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές. Με τον τρόπο αυτό ε, κατάλαβαν οι πολίτες ότι οι ανησυχίες τους ήταν βάσιμες. Τα αποτελέσματα της, ε, ε της ανάλυσης περιβαλλοντολογικής που έγινε μετά από ένα μήνα έδειξαν, έδειξαν πραγματικά ότι η, η κατάσταση του περιβάλλοντος ήταν πάρα πολύ άσχημη. Και τι έγινε τελικά, καλύφθηκε η δεξαμενή μέχρι ε, την μετακίνησή της. Αλλά μέχρι σήμερα δεν, ε, ε, δεν υπήρξε καμία άλλη προσπάθεια αποκατάστασης, δεν έγινε καμία ανάλυση για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται επιτόπου. Μετά από ε, κάποιες εργασίες ε, ε, σε, σε μια άλλη περιοχή δίπλα, φάνηκε ότι υπήρξαν διάφορες, υπήρχαν πάρα πολλά αποτελέσματα, όλα αυτά ήρθαν στο φως, περιμέναμε να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις, αλλά μέχρι σήμερα δεν έγινε τίποτα. Για να μην σας μιλήσω βεβαίως για τις καταγγελίες ε, που έγιναν ε, και, και για τις προσφυγές στη δικαιοσύνη ε, για, τις, για την παρουσία τοξικών αποβλήτων στην, ε, σας παραπέμπω και στην ε, δίκη Τεραμία η οποία έγινε σε μια ε, γειτονική περιοχή. Πάντως στις 17 Μαρτίου ε, ο δήμαρχος ε, του Μαριλιάνο της, ε, της πόλης μου ήρθε σε συμφωνία με, τον, με την Επιτροπή που ήταν υπεύθυνη για τα απόβλητα. Και ακριβώς εκεί υπήρξε κάποια προσπάθεια για να δούμε τι θα γίνει με τον προσωρινό χώρο αποθήκευσης. Όμως δεν καθορίζει, δεν υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα στην απόφαση αυτή. Και δεν φαίνεται τι θα γίνει με αυτά τα δισκία καυσίμου και ε, δεν υπάρχει στην ε, περιοχή μας, ε, παρά μόνο στην γειτονική περιοχή, καμία εγκατάσταση επεξεργασίας και πρέπει να σας πω ότι δεν έχουν χαρακτηριστεί οι χώροι. Και το πρώτο που θα πρέπει να γίνει είναι να χαρακτηριστούν οι χώροι αυτοί. Εξάλλου, όλα αυτά έχουν ανατεθεί ε, σε, σε κάποιες εταιρείε, ε, αλλά έχουν γίνει και κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές, όπως για παράδειγμα η εκπομπή Report, όπου έχουν, δει, όπου έχουν δείξει ότι αυτές οι εταιρείε δεν είναι ικανές να προβούν σε μετεγκατάσταση αυτών των χώρων. Από το 2004 μέχρι το 2004, η περιοχή μας, αλλά και η γειτονική δήμη, ε, ζήτησαν να γίνει ε, ανάλυση, δειγματοληπτική ανάλυση ε, του, του, στο γάλα των διαφόρων ζώων της περιοχής από μια, από μια κτηνιατρική επιτροπή και φάνηκε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος λόγω της διοξίνης. Επίση, στην Ατσέρα από το 2003 στο 2004 ε, υπήρξε σφαγή περίπου 5.000 ζώων και έγιναν ε, και διάφορες ε, αμβλώσεις επειδή τα, τα έμβρια αυτά ε, παρουσίαζαν πολλά, πολλά προβλήματα και τερατογενέσεις. Πρέπει να σας πω ότι ότι όσον αφορά την, παρουσία της διοξίνης υπάρχουν, έχουν, έχουν, έχουμε μεγάλη υπέρβαση των ορίων. Ένα χρόνο αργότερα πεθαίνει από, από, καρκίνος, από καρκίνο ο Ανδρέα Τζερλάντο, ο οποίος ήταν ε, ε, ε βοσκός ε, και στο αίμα του. Είχαμε επίσης υψηλή συγκέντρωση διοξίνης καθώς επίσης και βαρέα μέταλλα όπως ο μόλιβδος και το χρώμιο. Δεν υπήρξε λοιπόν ένα πρόγραμμα ε, βιολογικής ε, παρακολούθησης παρά μόνο το πολύ πρόσφατο χρονικό διάστημα ε, και με αποτέλεσμα οι κάτοικοι με δικά τους έξοδα να προβαίνουν σε ανάλυση και να φαίνεται ότι πραγματικά η διοξίνη βρίσκεται σε πολύ πιο υψηλά επίπεδα από τα αναμενόμενα. Πρέπει να σας πω ότι επειδή ε, συνεχίζονται οι γεωργικές δραστηριότητες στη χώρα μα, στην περιοχή μα μάλλον, πρέπει να γίνουν συγκεκριμένε έρευνε για να δούμε κατά πόσο τα προϊόντα αυτά τα οποία καλλιεργούμε και τα οποία καταναλώνουμε όλοι μα και τα οποία είπε και η συνάδελφο ότι έρχονται στο τραπέζι σα τελικά, να δούμε κατά πόσο υπάρχει σωστό έλεγχο και τι ακριβώ περιέχουν. Το 2008 ε, η, ε, η, η, κρατική αστυνομία στην έκθεση για την ζωομαφία ε, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου ε, λόγω ακριβώ. Ε, μία σαπάτη ε, που, ε, στην οποία εμπλέκονταν 649 ζώα, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο κλοπής και τα οποία προορίζονταν για σφαγή λόγω διοξίνης. φαίνεται λοιπόν ότι ενώ είχε γίνει ανάλυση στο, στο γάλα τους και είχε βρεθεί ότι, το, ότι υπήρξε μεγάλη ε, υπέρβαση των ορίων διοξίνης, τελικά τα ζώα αυτά αποτέλεσαν αντικείμενο ε, κλοπής. Από το Μάρτιο μέχρι το Μάρτιο 2009 ε, πρέπει να πω ότι είχαμε υπέρβαση των ορίων κατά 15 φορές και παραπάνω. Όλα αυτά τα φαινόμενα επαναλήφθηκαν και στη συνέχεια. Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται με την υγεία των πολιτών επιτόπου. Και τέλος, να σα πω το εξή. Εδώ δεν θα αναφέρω μία σειρά από σημεία τα οποία περιέχονται μέσα στο φάκελο και μέσα στα έγγραφα τα οποία σα δώσαμε. Πρέπει να σας πω ότι μετά από την ε, αναφορά μου, ε, πρέπει να σας πω ότι ε, είδαμε ότι ε, υπάρχει παρουσία ουσιών που είναι ιδιαίτερα τοξικές. Ξεκίνησε μία έρευνα σε δικαστικό επίπεδο από την εισαγγελία. Ε, προσπάθησα, προ, ε, να διαχωρίσουν ακριβώς την περιοχή στην οποία βρίσκονται οι, οι, οι, οι τοξικές αυτές ουσίες και να δούμε πώς θα γίνει αποκατάσταση και μεταφορά όλων αυτών των χώρων. Θέλω να πω με δύο λόγια ότι η ιστορία μας και το παρελθόν μας είναι γεμάτο τέτοια επεισόδια τα οποία δείχνουν πόσο σοβαρές είναι στο περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά, η γραφειοκρατική μηχανή είναι πάρα πολύ ε, αργή και αδρανή. Περνάνε τα χρόνια και δεν γίνεται τίποτα. Στο μεταξύ, βλέπουμε ότι έχουμε σοβαρέ περιπτώσει σοβαρών ασθενειών. Ε, καρκίνο, λευχαιμία κτλ. Σήμερα το πρωί μου αναφέρθηκε ε, ότι ένα θείο μου πέθανε από καρκίνο ένα χρόνο μετά από το θάνατο τη συζύγου του. Βεβαίω, εγώ δεν είμαι επιστήμονα, δεν ξέρω αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στα τοξικά απόβλητα, στην ρήπανση του περιβάλλοντο και Το γεγονό πάντω ότι, ότι βρίσκονται εκεί η, η, η, ρήπανση είναι ορατή, αλλά και η θάνατη είναι ορατή. Αυτό το οποίο λείπει είναι τα στοιχεία. Δηλαδή αυτό που θα μα επέτρεπε να καταλάβουμε το εύρο και τη διάσταση του προβλήματο. Ζητήσαμε αν είναι αλήθεια ή όχι το κατά πόσον ζούμε πράγματι στο τρίγωνο του θανάτου. Γιατί και αυτό ακόμα αμφισβητείται. Παρουσιάσαμε ένα φάκελο. Η, απο... η απάντηση ήταν ιδιαίτερα σαφή. Θέλουμε όμω βέβαιε απαντήσει ε, με, αυτή την... με, επιστημονική αυστηρότητα που οι πολιτικοί ζητούν από εμά. Εμά που δεν έχουμε τη δυνατότητα να, να δώσουμε τα στοιχεία. Ζητήσαμε από το Πανεπιστήμιο της Νάπολη να, ε, να μας κάνει μία ε, πρόβλεψη για το κόστος όσον αφορά τη χαρακτηριοποίηση του ε, της περιοχής μας. Ακούσαμε ένα ποσό, 60.000 ευρώ. Και όμως ακόμα τα πράγματα δεν έχουν προχωρήσει καθόλου. Αγαπητοί φίλοι, τι μπορούμε να κάνουμε για να αποδοθεί δικαιοσύνη, για να καταλάβουμε τελικά ε, την κατάσταση της περιοχής μας, την κατάσταση από άψη υγείας. Ε, οι θεσμοί μας δεν μας ακούνε, δεν παρεμβαίνουν όπως θα έπρεπε, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, αλλά και τους νόμους της χώρας μας. η δικαστική εξουσία με την καθυστέρησή της δεν μπορεί τελικά να αποκαταστήσει την αλήθεια οι πολιτικοί και τα αρμόδια όργανα υπεκφεύγουν δημιουργούν διάφορε έκτακτε επιτροπέ κτλ. Αλλά δεν μπορούν όλοι αυτοί να αντιμετωπίσουν και να λύσουν τα προβλήματα. Ο πολίτη έχει χάσει πια την εμπιστοσύνη του και ενώ καταπατούνται τα θεμελιώδη του δικαιώματα. Σήμερα ήρθαμε ενώπιον σα και, σας, ε, και εκπροσωπούμε τους πολίτες μας, ε, την, ε, την πατρίδα μας, την περιοχή μας. Υπό το φως όλων αυτών που σας καταγγέλουμε, ζητάμε να βοηθήσετε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς της χώρας μας, σε επιστημονικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο και σε οικονομικό επίπεδο. ερχόμαστε λοιπόν για να εκπροσωπήσουμε εδώ αυτούς που δεν έχουν φωνή, τους ασθενείς, τα παιδιά, αυτούς, τα, παιδιά για τα οποία να υπάρξει η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Σας ζητώ να παρέμβετε για να αποκατασταθεί η αλήθεια. Σας ζητώ να παρέμβετε για να αποκατασταθεί το δίκαιο, ε, η δικαιοσύνη. Αυτό ε, που διακηρύσει και το Ιταλικό Σύνταγμα, αλλά και, το Ευρωπαϊκό, ε, και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην υγεία, το δικαίωμα να ζει κανεί σε ένα καθαρό περιβάλλον, σε ένα υγιεινό περιβάλλον. Αναφέρε τα δικαιώματα, τα οποία αναγνωρίζονται από όλα τα δίκαια και από, όλους, και από όλες τις χάρτες θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σας καλώ λοιπόν να υπάρξει μια πραγματική επιτροπή, ε, όχι στα χαρτιά, αλλά ε, ε, που να δει με τα δικά σας μάτια. ε, δεν αρκούν οι τιμωρίες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δοθεί εντολή σε έναν ευρωπαϊκό φορέα, όχι Ιταλό, αλλά διεθνή, για να παρακολουθηθεί η συγκεκριμένη κατάσταση επιτόπου, να χαρακτηριστεί η συγκεκριμένη περιοχή, να παρακολουθηθεί η κατάσταση υγείας των πολιτών με συγκεκριμένε έρευνε. Σα ευχαριστώ για την υπομονή σα. Σα ευχαριστώ εξ εξ των πολιτών του Μαριλιάνο ε, και τη ευρύτερη περιοχή. Σα ευχαριστώ και σα εύχομαι ε, να συνεχίσετε την εργασία σα με τον καλύτερο τρόπο. Σα ευχαριστώ όλους σα. Βεβαίω αυτά τα πράγματα είναι ε, τρομερά και ξέρετε όλοι ότι εγώ δίνω μεγάλη σοβαρότητα στα πράγματα αυτά. Ξέρω ότι είπατε να μην είναι κάποιο Ιταλό που θα ασχοληθεί με όλα αυτά. Εγώ ω Ιταλίδα θέλω να βοηθήσω έτσι ώστε να αλλάξει η εικόνα, έστω στο ελάχιστο, όσον αφορά δηλαδή την πολιτική εκπροσώπηση και του πολιτικού γενικότερα. Λοιπόν, τι σα έλαχε να είμαι εγώ πρόεδρο τη Επιτροπή, που είμαι Ιταλίδα και ζητώ συγγνώμη για το αστείο μου. Ε, θέλω να πω ότι ω Ιταλίδα όμω θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να ακουστούν οι ανάγκε σα και αυτά τα οποία ζητάτε σε ζητώ συγγνώμη. Ε, α, έχουμε και άλλον έναν. Το Μάση Εσπόζητο. Για την 347-2008. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω ε, την Επιτροπή σας που μας δίνει τη δυνατότητα να έρθουμε εδώ και να ε, εκπροσωπήσουμε τις ε, περιοχές μας. Εγώ ε, σας παραπέμπω στα έγγραφα που έχουμε καταθέσει ε, στο φάκελό σας ε, σε όλα αυτά τα οποία καταθέσαμε με τα γεγονότα τα τότε, τότε η κυβέρνηση πρώτη, που είχε αναφερθεί σε αυτή την απόφαση για την εγκατάσταση αποτέφρωσης. Και ε, βεβαίω θα ήθελα να πω εδώ ότι ε, μιλάμε για την παραβίαση μια σειρά από κοινοτικών οδηγιών. Και ε, παρακλίνοντα από την από, από την περιβαλλοντική αξιολόγηση του Φεβρουαρίου 2005 με, με βάση ε, την οποία ε, αναφερόταν ε, το, το Υπουργικό Διάταγμα του 1998 που προέβλεπε την, τη δυνατότητα να αποτελούν αντικείμενα αποτέφρωσης μόνο συγκεκριμένα απόβλητα. Δεν μπορούσαν δηλαδή να καίγονται όλο κάθε είδους απόβλητα. Εμείς είδαμε ότι μέσα από τη, με την πάροδο του χρόνου είχαμε παραβίαση πολλών οδηγιών και κυρίως το 2001 77 που αναφερόταν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, τη 2076 ε, για τα απόβλητα και την την οδηγία 85337 που μιλούσε για την περιβαλλοντική αξιολόγηση διαφόρων δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Λοιπόν, όσον αφορά ε, την απάντηση που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που για σας τα μέλη του Κοινοβουλίου αποτελεί μία γνωμοδότηση στην οποία και εμείς θα θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο εξή. και ελπίζω ε, να μην ε, ε, να μην σταματήσετε τις προσπάθειές τα σήμερα και να καταλάβετε τι ακριβώς πιστεύουν και οι θεσμοί αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής. Λοιπόν, να σας πω συγκεκριμένα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ουσία έδωσε διευκρινήσεις που δεν καλύπτουν όμως διεξοδικά το ζήτημα. Είναι σωστό, είναι αλήθεια ότι η Επιτροπή αρχικά αναγνώρισε την μη ορθή εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο ε, για τα απόβλητα 2006-12 ΕΟΚ ε, και, και αναγνωρίζει ότι υπάρχει διαδικασία, πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία παράβασης, ε, παραβίασης κατά της Ιταλίας ε, και αναγνωρίζει την έλλειψη των υποδομών για τη διαχείριση των, αποβλητών, των αποβλήτων, δεν απάντησε συγκεκριμένα. Απάντησε μόνο γενικά και δεν απάντησε στις ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν αρκείται στο να παρατηρεί την κατάσταση. Πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση στην καμπάνια συγκεκριμένα εξακολουθεί να είναι η ίδια ε, εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η έκτακτη επιτροπή ε, παρακολούθηση τη διαχείριση των αποβλήτων που ξεκίνησε το 1994. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει τελικά και μετά από τόσα χρόνια εξακολουθεί στο όνομα μια έκτακτη ανάγκη ε, να υπάρχει παρέκκληση από όλη την ε, νομοθεσία που αφορά το θέμα, από την ε, προϋπόθεση ύπαρξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων κτλ. Έχουμε λοιπόν παραβίαση μια σειρά από νομοθεσιών που αναφέρουμε ε, και στην αναφορά και πρέπει να πω στη συνέχεια ότι με την ε, κυβέρνηση Μπερλουσκόνη Ε, Ακριβώ αυτά τα διατάγματα τα οποία επιτρέπουν, ήρθαν, στην επιφάνεια τα διατάγματα τα οποία επιτρέπουν ε, την αποτέφρωση όλων των αποβλήτων χωρί καμία περιβαλλοντική αξιολόγηση και ε, μπορούμε πλέον να έχουμε εκ νέου χρησιμοποίηση τη ενέργεια που προέρχεται από αυτού του αποτεφρωτέ, από τι εγκαταστάσει αποτέφρωση. Έχουμε ταυτόχρονα στρατιωτικοποίηση τη ε, περιοχή. Δηλαδή, εδώ έχουμε παρακολούθηση ε, και έλεγχο των εγκαταστάσεων από το στρατό. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε παραβίαση κάθε αρχής δικαίου και μιλάμε 15 χρόνια μετά από την εμφάνιση των έκτακτων περιστάσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν δεν έχει απαντήσει διεξοδικά, ε, δεν υπάρχει οριστική διαχείριση του αποτεφρωτή, ε, καίγονται ανεξαρτήτως τα απόβλητα, ε, δεν γίνεται ε, ε, ε, ε διαλογή στην συγκομιδή και στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Στην καμπάνια πρέπει να σας πω ότι δεν έχει ξεκινήσει καν η, η διαλογή ε, ε, όπως σας είπα καίγονται ε, αδιακρίτως όλα τα απόβλητα, εξακολουθούν να είναι πολύ μεγάλες οι ανησυχίες στην περιοχή αυτή. Έχουμε μεγάλες περιπτώσεις τερατογενέσεων και, και κρουσμάτων καρκίνου και αυτό έγινε, επιβεβαιώθηκε και από μια έκτακτη επιτροπή με έναν έκτακτο επίτροπο Μπερτολάζο και επιβεβαιώθηκαν τα στοιχεία αυτά και από την Παγκόσμιο Οργάνωση Υγείας και από άλλους οργανισμούς που αναγνώρισαν την σοβαρή κατάσταση. Λοιπόν, τα πρώτα στοιχεία ε, επιβεβαιώνουν ε, τις ανησυχίες μας. Ε, η Περιφερειακή Αρχή για την Προστασία του Περιβάλλοντος έδωσε τα στοιχεία σε ένα παρατηρητήριο και ε, φαίνεται δεν μπορεί να κάνει άλλο παρά να αναγνωρίσει παρόλες τις προσπάθειες προς την αντίθετη κατεύθυνση ότι μέσα σε 8 μήνες από τις 26 Μαρτίου ε, του 2009 μέχρι σήμερα ε, παρατηρήθηκε, ε, παρατηρήθηκαν συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα τοξικών ουσιών 100 φορές πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Και επίσης να σας πω, εντάξει εμείς έχουμε πολλές ιδιομορφίες στην Ιταλία ε, και πρέπει να σας πω ότι ε, ο, ο πρόεδρος αυτής της αρχής που παρακολουθεί την κατάσταση στο περιβάλλον είναι πρώην πρόεδρος της Επιτροπής ε, που είχε αποφασίσει για τον αποτεφρωτή. Δηλαδή εδώ μιλάμε για μια συνεχή έλλειψη προστασίας των κατοίκων. Και εκ μέρους της Επιτροπής δεν υπήρξε καμία διευκρίνηση όσον αφορά όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι σαφές ότι στην περιοχή μας οι πολίτε είναι αυτοί που θα πληρώσουν το κόστο ε, μέσω του λογαριασμού τη ΔΕΗ. Δεν γίνεται καμία διάκριση ε, ε, ανάμεσα στις, στο κατά πόσο έχουμε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια ή άλλη μορφή ενέργεια. έτσι κι οι καταναλωτέ τα πληρώνουν όλα. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι ε, αυτή τη στιγμή ε, ενώ, ε, ενώ μιλάμε ε, για επιδότηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εδώ μιλάμε στην ουσία για επιδότηση ενέργειας που έρχεται από τους αποτεφρωτές αυτές που όμως δεν είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μιλάμε λοιπόν ε, για μείωση των ε, κονδυλίων και των επιδοτήσεων για την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Είναι τρομερέ οι ανησυχίε και για τη ρήπανση του περιβάλλοντο, ε, γιατί έχουμε σημαντικέ εκπομπέ τοξικών ουσιών και μιλάμε για μια περίοδο τη παραμονή τη Κοπεχάγη όπου θα ζητηθούν όλα αυτά τα θέματα τα τόσο σοβαρά και που αφορούν το κλίμα και την αλλαγή του κλίματος. Θέλουμε λοιπόν σημαντικές απαντήσεις και διαφάνεια. Δεν είδαμε να υλοποιείται κανένα σχέδιο μέχρι στιγμή και τελειώνω βεβαίω εδώ και, θα ήθε... και αντιλαμβάνομαι ότι το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ δύσκολο να εξηγηθεί ε, και να το εξηγήσω και σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Ε, σας παραπέμπω λοιπόν στα αντίστοιχα έγγραφα. Νομίζω ότι θα πρέπει να, να... γίνει παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, γιατί πρέπει να σας πω ότι μέσα στις παρατηρήσεις της Επιτροπής φάνηκε ότι υπάρχει διαδικασία παραβίασης και καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί ακριβώς ε, δεν υπάρχει ε, καμία πολιτική επιτόπου προς την ορθή κατεύθυνση. Ζητούμε λοιπόν ε, να υπάρξει απόφαση του, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το θέμα της υποδομής για τη διαχείριση των αποβλήτων. Δεν έχει λυθεί τίποτα προς την κατεύθυνση αυτή. δεν ακολουθήθηκε η αρχή της προφύλαξης, με βάση την οποία δεν πρέπει να ε, ρηψοκινδυνεύουμε καθόλου ότι μπορούμε να κάνουμε αλλιώ και να περιμένουμε λοιπόν να ανασταλούν όλα αυτά μέχρι να έχουμε την οριστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Να, υπάρξουν, λοιπόν, ε, να υπάρξει μια πραγματική πολιτική διάθεση των αποβλήτων σε κάθε στάδιο. Διότι διαφορετικά δεν παροβιάζουμε μόνο την παλιά οδηγία του 2006, αλλά και την καινούργια οδηγία τη κοινότητα ε, επί του θέματο. Ζητάμε λοιπόν η Επιτροπή Αναφορών και, και σα ευχαριστώ βεβαίω για άλλη μια φορά για την προσοχή σα και για την υπομονή σα. Ζητούμε να, να αποστείλετε σημείωμα προ την ε, Ιταλική κυβέρνηση για όλε αυτέ τι παραβιάσει και καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει κάθε μέτρο έτσι ώστε να απαιτήσει ε, τον, την εκπλήρωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ή να δοθεί κάποια ε, ε, απάντηση λογικοφανής που μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί. Ο κύριος Βιτσέντσο Μάρμαρα είναι και αυτός παρόν. Όχι. Ε, allora, a questo punto darei la Τώρα στο σημείο αυτό να δώσουμε το λόγο στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Grazie Σας ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους αναφέροντες που ήρθαν εδώ σήμερα για άλλη μια φορά για να παρουσιάσουν τις, ε, και να εξηγήσουν τις αναφορές τους. Και θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε, να σας ζητήσω να μου επιτρέψετε να απαντήσω συνολικά στις διάφορες αναφορές που αφορούν τα απόβλητα στην καμπάνια. Ε, δηλαδή και στα δύο σημεία, 12 και 13 της ημερήσιας διάταξης. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή συνειδητοποιεί απόλυτα το γεγονός ότι στην καμπάνια τα τελευταία χρόνια επήλθαν όλες αυτές οι επανειλημμένες παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου όσον αφορά τα θέματα περιβάλλοντος. Τα προβλήματα τα οποία αναφέρθηκαν μέσα στις αναφορές και που επαναλήφθηκαν και σήμερα μέσα από τις διάφορες προφορικές παρεμβάσεις και που, μίλησαν για, και που μιλούν τελικά για εγκατάλειψη των ε, αποβλήτων στο δρόμο, κατά μήκο του δρόμου, ή ε, στους διάφορους χώρους αποθήκευσης κτλ. Όλα αυτά στην ουσία και κατά την άποψη Επιτροπής δείχνουν ένα θεμελιώδες πρόβλημα. Ποιο της έλλειψης στην Καπανία ενός πραγματικού δικτύου υποδομών για την διαχείριση ε, και την διάθεση των αποβλήτων. Κατά την άποψή μας, μόνο εξασφαλίζοντας την παρουσία ενός επαρκούς αριθμού ε, εγκαταστάσεων ε, επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων, μόνο τότε η κατάσταση στην Καπανία θα μπορέσει να ομαλοποιηθεί και μόνο χάρη σε ένα σύστημα διαχείρισης και επεξεργασίας των αποβλήτων, το οποίο ε, ε, να είναι ένα πραγματικό σύστημα ε, διάθεσης, μόνο τότε θα μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι αποφεύγονται αυτοί οι κίνδυνοι και οι σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον. Άρα μόνο τότε θα μπορέσουμε να έχουμε την εγγύηση εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας. Να σας πω λοιπόν αυτό το οποίο έκανε τα, τα τελευταία αυτά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρόλο που κατά την άποψη των ε, αναφερόντων δεν ήταν αρκετά. Όταν ε, ενημερωθήκαμε για την κρίση για τα απόβλητα την άνοιξη του 2007, αμέσως ε, ξεκινήσαμε διαδικασία επιπαραβάση. Και ε, είπαμε στην ε, Ιταλία ακριβώ αυτό, ότι δεν υπάρχει ε, το δίκτυο υποδομή για τη διάθεση και την επεξεργασία αποβλήτων με του όλου του κινδύνου που συνεπάγεται κάτι τέτοιο για τη δημόσια υγεία και για το περιβάλλον. Στείλαμε λοιπόν την πρώτη προειδοποιητική αποστολή και ακολούθησε μία σειρά από συναντήσεις των υπηρεσιών μας με τις αρμόδιες αρχές στην Ιταλία. Ορισμένες συναντήσεις διεξήχθησαν επιτόπου. Ήδη από τον Ιούλιο του 2007, μία αντιπροσωπεία της Επιτροπής πραγματοποίησε μία πρώτη επιτόπου επίσκεψη. Και τότε φάνηκε το πρόβλημα σε όλο το μεγαλείο. Ε, αποβλήτων που συγκεντρώνονται στους δρόμους και πολυάριθμοι ε, χώροι που φαίνονταν και από το αεροπλάνο την ώρα που προσγειωνόταν, ε, χώροι αποθήκευσης. Η ανάλυση λοιπόν της Επιτροπής έδειξε ότι η ρίζα του προβλήματος είναι η ανεπαρκής ικανότητα διάθεσης των αποβλήτων σε περιφερειακό επίπεδο. Η παραγωγή αποβλήτων στην καμπάνια υπερβαίνει τις 7.000 τόνους ημερησίως και τότε, δηλαδή τον Ιούλιο του 2007, η ικανότητα διάθεσης στην περιοχή ήταν μηδενική σχεδόν. Ε, οι χώροι υγειονομικής ταφής που υπήρχαν ε, είχαν σχεδόν ε, εξαντληθεί ως προς τη δυνατότητά τους. Η κατασκευή νέων υποδομών συμπεριλαμβάνοντας και τον αποτεφρωτή του Ατσέρα είχαν καθυστερήσει ιδιαίτερα. Το περιφερειακό σχέδιο για τα απόβλητα δεν είχε υλοποιηθεί. Ήδη υπήρχαν στοιχεία τα οποία καταδείκνυαν ότι η κρίση των αποβλήτων αποτελούσε γόνιμο έδαφος για το οργανωμένο έγκλημα. Ε, και για παράνομες επιχειρήσεις διάθεσης αποβλήτων. Ο Ιταλικός τύπος υπενθύμησε επανειλημμένα ε, και έφερε στο φως πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το ε, οργανωμένο έγκλημα εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται την περιοχή για την παράνομη διάθεση ακόμα και τοξικών αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων δεδομένης ε, της διάρκειας της κρίσης, η διαδικασία παραβάση που ξεκίνησε η Επιτροπή προχώρησε. Και το Μάιο του 2008 αποφασίσαμε ε, να ε, προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτή τη στιγμή η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της αναμονής της απόφασης. Και πιστεύω ότι η απόφαση του δικαστηρίου θα έρθει μέσα στους προσοχείς δύο ή τρεις μήνες. Ακριβώς για αυτό το γεγονός δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο σήμερα και να τοποθετώ περισσότερο για αυτές τις αναφορές που γιατί όπως σας είπα η υπόθεση κρεμεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Θα ήθελα όμως να επιβεβαιώσω το ότι ε, η υλοποίηση ενός επαρκού δικτύου υποδομής ε, ε, για τη διάθεση και την επεξεργασία των αποβλήτων βεβαίως είναι στοιχειώδης και βασική, αλλά θα αποτελέσει μόνο το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση της ομαλότητας στην περιοχή. Η περιοχή της Καμπάνιας θα πρέπει να εφοδιαστεί με μια ολοκληρωμένη στρατηγική διάθεση των αποβλήτων μέσα από την ορθή εφαρμογή της υφιστάμενης κοινοτικής νομοθεσίας και ε, μέσα από την ορθή πρόβλεψη ε, διαφόρων ε, συστημάτων όπως διαφοροποιημένης και χωριστής περισυλλογής, ανακύκλωσης βεβαίως και για να μην σας αναφέρω το γεγονός ότι πήγει απόλυτα να υπάρξει σημαντική μείωση της μάζας των αποβλήτων. Και να σας πω και το εξής και να κάνω ορισμένε παρατηρήσεις ε, γενικότερης φύσεως. Από τη μια η Επιτροπή ε, ξεκίνησε τη διαδικασία κατά της Ιταλίας για το θέμα αυτό της κρίσης για τα απόβλητα στην Καμπανία και αυτό είναι αλήθεια. Από την άλλη, λοιπόν, η λιμένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθύμησε στις Ιταλικές Αρχές την ανάγκη σεβασμού του, της κοινοτικής νομοθεσίας και της λήψης των επαρκών μέτρων εξόδου από την κρίση τόσο όσον αφορά τι ε, κανονιστικές διατάξεις σε, περι, σε περιπτώσεις, έκτακτη ανάγκη και εδώ σας παραπέμπω ε, στις ε, ε επανειλημμένες επαφές που είχαν οι υπηρεσίε μας με, με τις αρχέ Αρχές ε, για την ε, μετατροπή σε νόμο του διατάγματος 90-22 ε, ε, του 2008 ε, ε, για τους αποτεφρωτέ κτλ. Δηλαδή, οι υπηρεσίε τη Επιτροπής παρενέβησαν προληπτικά για να μην υπάρξει δηλαδή περαιτέρω παραβίαση του κοινοτικού δικαίου μέσα από αυτά τα έκτακτα μέτρα. Αυτή η δράση ε, έγινε και με ανταλλαγή επιστολών, αλλά και με συγκεκριμένε επιτόπου επαφέ σε επίπεδο τεχνικών εμπειρογνωμόνων. Οι ιταλικέ αρχέ επανειλημμένα εξέφρασαν τη δέσμευσή του απέναντι στην ορθή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Επομένω, η Επιτροπή μέχρι σήμερα δεν έχει λόγο να θεωρεί ότι οι νέε εγκαταστάσει διάθεση, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο στάδιο ε, τη ε, ε, κατασκευή στην περιοχή, δεν θα σέβονται την κοινοτική νομοθεσία. Εξάλλου, δεν πρέπει να σα δημιουργήσει έκπληξη το γεγονό ότι οι καταγγελίε ε, ε, και οι προσφυγέ προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πολύ πολυάριθμες ε, η αντίδραση των κατοίκων στην κατασκευή εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων είναι κάτι το κατανοητό. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για μια κατάσταση όπως αυτή στην περιοχή της Καμπανίας. Γιατί εκεί έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα δυσπιστίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε με πολύ μεγάλη προσοχή όλες αυτές τις καταγγελίες που μας έγιναν και όπου υπήρξε ανάγκη ζητήσαμε διευκρινήσεις από τις τελικές αρχές. Όσον αφορά τώρα τους νέους χώρους διάθεσης αποβλήτων, στην καμπανία, μέχρι στιγμής δεν κατέστη αναγκαία ανάληψη δράσης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πέραν βεβαίως ε, των διευκρινιστικών ερωτήσεων. Σε σχέση με το θέμα αυτό, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ποια είναι τα όρια ε, της δράσης της Επιτροπής και ε, ποια είναι τα προνόμια των κρατών μελών. Η Επιτροπή δεν μπορεί ούτε πρέπει να υποκαθιστά τα κράτη-μέλη στις αποφάσεις τους για τις ε, νέες εγκαταστάσεις διάθεσης. Εφόσον ε, τηρείται το κοινοτικό δίκαιο, οι αποφάσεις των εθνικών αρχών ε, όσον αφορά ε, την κατασκευή νέων χώρων υγειονομικής ταφής ή εγκαταστάσεων αποτέφρωσης, δεν έχουμε εμεί κανένα λόγο σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να... θα ήθελα να κάνω τώρα μία διευκρίνηση όσον αφορά την τελευταία αυτή παρέμβαση και που αφορούσε την ατσέρα και τη συγκεκριμένη αναφορά. Όσον αφορά την αντίστοιχη οδηγία, πρέπει να πω ότι η οδηγία αυτή δεν αναφέρει ότι οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εξετάσουν άλλες εναλλακτικές λύσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Εξάλλου, η συγκεκριμένη οδηγία προβλέπει ότι οι αρμόδιες αρχές όταν δίνουν την άδεια σε ένα σχέδιο το οποίο υπόκειται στην οδηγία αυτή, λαμβάνουν υπόψη ε, τις ε, μελέτες ε, επιπτώσεων στο περιβάλλον, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, καθώς επίσης και τη διαβούλευση με τις περιοδολικές αρχές. Όμως θα πρέπει να διευκρινιστεί και αυτή η διευκρίνηση είναι ουσιώδους σημασίας ότι αυτή η οδηγία δεν προβλέπει ότι όλα αυτά είναι δεσμευτικά. Το γεγονός ότι ορισμένες από τις ε, ε αποφάσεις της ε, Ιταλικής Επιτροπής ε, για τη συγκεκριμένη οδηγία δεν έγιναν σεβαστές όσον αφορά την οριστική επιλογή του χώρου και την πραγματοποίηση του τόπου, αυτό δεν αποτελεί παραβίαση της συγκεκριμένη οδηγίας. Αν προκύψει ανάγκη, θα ζητήσω και από τους συναδέλφους να παρέμβουν σε σχέση με την Οδηγία 2001 του 77. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και στο συγγνώμη γιατί μακρηγόρησα. Εγώ σας ευχαριστώ. Βεβαίως, αλλά ήταν απαραίτητο. Έπρεπε να αναφερθούν όλα αυτά τα στοιχεία. Όμως έχουμε μόλις 14 λεπτά στη διάθεσή μας. Προσπάθησα να ζητήσω λίγο περισσότερο χρόνο. Έχω πολλούς συναδέλφου που ζητούν το λόγο. Σας ζητώ να είστε σύντομοι για να μπορέσουμε να κλείσουμε το θέμα. Και ίσως να ακούσουμε και τους ε, άλλους συναδέλφους της Επιτροπής που ενδεχομένως να έχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις. Επιτρέψτε μου, ε, έστω και καθυστερημένα, να καλωσορίσω την κυρία Φρασόνη που είναι, κοντά, που είναι μαζί μας σήμερα και να δώσω πρώτο λόγο στην κυρία Όκεν. Øh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους αναφέροντες γιατί έχουν κάνει πολλή δουλειά και θέλω να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί έδωσε μία αρκετά εκτεταμένη απάντηση. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λυπάμαι, αλλά είναι τμήμα του προβλήματος και όχι τμήμα της λύσης. Γιατί δεν έχουν γίνει αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει. Μπορεί να ε, συζητάμε πολλά πράγματα, αλλά δεν έχει ληφθεί δράση. Και εδώ έχουμε ένα τεράστιο πολιτικό σκάνδαλο. Είναι κάτι το οποίο χρόνια τώρα διαρκεί και περιγράφεται και στον τύπο στη Δανία. Και χαίρομαι που είπε η πρόεδρο ότι θα αντιμετωπίσουμε το θέμα και θα παραμείνουν ανοιχτέ οι αναφορές και όλα αυτά. Πρέπει όμω να δούμε ότι στην πράξη δεν έχει γίνει τίποτα. και βλέπουμε ότι δίνονται εγκρίσει, παραδείγματο χάρη, για την κατασκευή από τεφροτήρα. Ενώ αγνοούνται όλε οι διατάξει των οδηγιών σχετικά με τους αποτεφρωτήρες. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι επίγον το θέμα και να πρέπει να κατασκευαστεί ένα αποτεφρωτήρα, αλλά δεν μπορεί να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε ένα κίνδυνο δημιουργώντα ένα νέο κίνδυνο. Ένας αποτεφρωτήρας δημιουργεί ρήπανση και γνωρίζω τους κίνδυνου από την καύση χημικών και από τα όσα διαβάζουμε στι εφημερίδε στη Δανία. Πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε οι προποθέσει. και η οδηγία για τα απόβλητα φαίνεται να αγνοείται, να παραμερίζεται. Πρέπει να δούμε ε, τι πρέπει να γίνει σωστά. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Λέμε ότι υπάρχουν τα θέματα των ανανεώσιμων ε, πηγών ενέργειας, ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, κρατικές ενισχύσεις. Τι θα γίνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ιταλία. Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει να στείλουμε μια αντιπροσωπεία για να μιλήσει με τους ανθρώπους επιτόπου. Πρέπει να βρεθεί μια λύση για αυτή την υπόθεση. και δεν είναι ένα περιορισμένο θέμα, νομίζω ότι είναι ένα ευρύτατο θέμα και είναι κάτι που μας αφορά όλους. Εξάλλου την Ιταλία όλοι την αγαπάμε και αυτές τις περιοχές στην Καμπανία όλοι τις αγαπάμε. Να μην αφήσουμε να προσθέσετε ρήπανση στη ρήπανση που ήδη υπάρχει. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Ριβελίνη, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σα πω ότι εγώ είμαι από αυτή την περιοχή και πρέπει να σα πω ότι αντιμετωπίζω τρομερέ δυσκολίε Γιατί είμαι πολίτη τη περιοχή και είμαι δίπλα ακόμα ε, και σε αυτού που υπέβαλαν την, ανα, την αναφορά και βρίσκονται εδώ, ε, σε αυτή την αίθουσα, ε, όταν, μιλούσαν έκανε διαμαρτυρία για το ταβέρνα Ντελρέ. Ε, πρέπει να σας πω ότι ήμουν ε, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος σε, περιφερειακό επίπεδο και, και συζήτησα αυτό το περιφερειακό σχέδιο για τα απόβλητα που εγκρίθηκαν, που εγκρίθηκε καθυστερημένα. Σήμερα είμαι Ευρωπαίο πολίτη, είμαι μέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με αυτή τη στιγμή πρέπει να σα πω ότι αγανακτώ αν ακούω ότι ε, βλέπω ότι εξακολουθούμε να φλιαρούμε χωρί να λέμε τα πράγματα με το όνομά του και χωρί να ε, τολμάμε να αντιμετωπίζουμε ε, την πραγματικότητα. Και ποια είναι η αλήθεια, ότι από το 2001 στο 2008 και πάλι καλά που ήρθε ο Μπερτολάσο και ευτυχώ που ήρθε ο Μπερλουσκόνη υπήρξαν περιφερειακές πολιτικές ε, επιζήμιες, ε, ολέθριε. Ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης ε, και βρισκόμουν στο κοινοβούλιο όταν είχαμε τα απόβλητα κατά μεσή στο δρόμο, όταν γίνονταν αυτές οι αναλύσεις που έδειχναν ε, αύξηση των καρκίνων κατά 14% στην περιοχή μας. Ε, όταν ε, ε, το δικό μου το κόμμα ήταν παρόν ακριβώς στην περιοχή μου όταν είδαμε ότι από τις 30 γυναίκες και 30 είχαν όγκο. Και να ακούω λοιπόν αυτές τις φλιαρίες. Γιατί το λέω, φλιαρίες. για τα απόβλητα, μηδενικά απόβλητα, τέτοιες βλακίες. Εγώ τι να σας πω. Η αλήθεια, ποια είναι η αλήθεια. Δεν δέχομαι ούτε αυτό που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να στείλουμε μια επιτροπή εξεταστική για να καταλάβει το πώς το 2008, πώς το καλό, χωρίς κανένα προγραμματισμό, έκλεισαν οι χωματερές, οι, χώροι υγειονομικής ταφής, αφήνοντας τους κατοίκους της περιοχής στις αρρώστιες και στα απόβλητα σκουπίδια μέσα στο δρόμο. Πώς έγινε αυτά τα κόμματα της αριστεράς, οι πράσινοι, μέσα στο κοινοβούλιο φώναζαν απόβλητα μηδέν και απ' την άλλη κάτι και υπέφεραν και αναρωτιέμαι. Και γι' αυτό δεν είμαι, δεν συμφωνώ με αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δύο χρόνια πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήγε επί Έκανε παλήθευση. Τι έγινε. Ποιες ήταν οι έρευνες, οι εκθέσεις που απεστάλησαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε αυτούς τους ε, πολίτες στην Καπανία που ε, αντιμετωπίζουν τρομερές ασθένειες. Κοιτάξτε τι να σας πω, με μία τροπολογία μου καταφέραμε να δώσουμε 500.000 ευρώ για να καταλάβουμε τα επίπεδα διοξίνης στο αίμα των πολιτών στο ταβέρνα Ντερρέ. Έκανα αγώνα και τελικά τα καταφέραμε όλα αυτά. Λοιπόν, αυτή η επιτροπή καθοδηγούμενη από έναν Ιταλό, τον Πρόντι. Τι, σε τι αποτέλεσμα ε, μας οδήγησε. Και σήμερα είμαι μέλο του Κοινοβουλίου τη Ευρώπη και είμαι Ευρωπαίος πολίτης έτσι και ρωτώ. Η Ευρώπη τελικά θέλει ε, να, ε, να δείξουμε τι έγινε σε αυτά τα χρόνια όταν τα σκουπίδια πουλιόντουσαν σαν χρυσάφι ε, στους Γερμανούς. Και αυτή η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει τελικά να αντιληφθεί τη ζημιά στο περιβάλλον, στην καμπάνια. Αγαπητοί φίλοι, που είναι η πατρίδα της Μεγάλης Ελλάδας, που είναι το λίκνο ε, του πολιτισμού. Τα γεωργικά μας προϊόντα είναι τα καλύτερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ποιος θα, θα τα πληρώσει όλα αυτά. Ποιος θα, θα, θα αποζημιώσει τη γη μας ε, για αυτές τις ζημιές. Το ξαναλέω. Ευχαριστώ τους πολίτες που ήρθαν εδώ, γιατί δείχνουν ότι εδώ υπάρχει η κοινωνία των πολιτών και με μια στάση που είναι σίγουρα θετική. Αλλά τελικά θα πρέπει να ανοίξει, ε, να υπάρξει μια πραγματική εξεταστική επιτροπή ε, για να καταγγείλει αυτό το οποίο έγινε το 2000-2008. Αυτό είναι το ένα. Να ξεκινήσει μια ευρωπαϊκή πολιτική. Γιατί Κοιτάξτε, όπω ένα μεγάλο σεισμό, μια μεγάλη φυσική καταστροφή, ένα κατακλυσμό, αυτά έχουν επιπτώσει σε όλου. Απαιτούνται λοιπόν κονδύλια. Θέλει προσοχή η συγκεκριμένη περιοχή. Και τέλο, ζητώ από την Επιτροπή να κάνει κάτι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και οι διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Γιατί και με τον τρόπο αυτό θα δώσουμε στους πολίτες, σε αυτούς τους πολίτες που τιμωρήθηκαν, τη δυνατότητα να ζητήσουν αποζημίωση και να ζητήσουν αποκατάσταση των δικαιωμάτων τους. Ευχαριστώ κύριε Μποσινάρου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εντάξει, εδώ δεν μιλάμε ούτε για την Ασία ούτε για την Αφρική. Μιλάμε για ένα ιδρυτικό μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καθαρά ευρωπαϊκό θέμα και αφορά μια συνεχιζόμενη παραβίαση ευρωπαϊκών κανόνων και νομοθεσίας. Τελεία. Εγώ προτείνω να οργανώσουμε μία αποστολή διερευνητική και να έχουμε πριν από την αποστολή ενημερωθεί επισήμως, να έχουμε και την επίσημη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί ακούστηκαν ωραίες ιδέες για το τι πρέπει να γίνει στην Ιταλία, αλλά τίποτα συγκεκριμένο δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Και θέλουμε και την επίσημη θέση της Ιταλικής κυβέρνησης και με τις πληροφορίες αυτές του χρόνου την Άνοιξη να πάμε στην Ιταλία, να πάει μια αποστολή από την Επιτροπή μας γιατί είναι τόσο πολλές κοινότητες και τόσο πολλοί πολίτες που αξίζουν πραγματικά τη βοήθειά μας. Ευχαριστώ. Μάρκες. Κυρία Μάρκες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προφανώς είναι μια κατάσταση δύσκολη και επικίνδυνη και επίγουσα. Και συμφωνώ με τον κύριο Μποσινάρο και όπως ήδη ελέγχθηκε από άλλου συναδέλφου, πρέπει να διοργανώσουμε μια διερευνητική αποστολή και να προσπαθήσουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Έχω αρκετέ ερωτήσεις. Συμφωνώ με κάποιον προηγούμενο μιλητή που είπε ότι λέγονται πολλά, αλλά μένουμε στα λόγια, δεν βλέπουμε έργα. Γι' αυτό έχω και εγώ πολλά ερωτηματικά. Ακούμε ότι η Επιτροπή παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την κατάσταση στην Καμπανία και τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν ή προγραμματίζουν οι Ιταλικές αρχές και προσπαθεί να δει τι άλλο μπορεί να γίνει για να επιληθεί και η επίγουσα κατάσταση και η διαρθρωτική κατάσταση έχουν μια γενική εικόνα των όσων συμβαίνουν. Παρακολουθεί αρκετά προσεκτικά την κατάσταση η Επιτροπή. Εγώ θα ήθελα να δω ποια είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί, τα μέτρα που έχουν ήδη προγραμματίσει οι Ιταλικές Αρχές. Άλλη ερώτηση. Ακούσαμε ότι δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αξιολογήσει τους κινδύνους που έχουν σχέση με εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων. Δεν μπορεί να παρέμβει η Επιτροπή εφόσον οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία. Αλλά έχουν ληφθεί αποφάσεις με βάση την κοινοτική νομοθεσία. Φαίνεται ότι διαφέρουν τα πράγματα στη θεωρία και στην πράξη. Μπορεί οι αποφάσει να είναι συμβατέ με την νομοθεσία, αλλά η εκτέλεση του η υλοποίηση των αποφάσεων δεν είναι συμβατή με την κοινωτική νομοθεσία. Και έχω και κάποια πιο πρακτικά ερωτήματα. Αν είναι όντω τόσο επίγουσα η κατάσταση και από ό,τι φαίνεται και από την αξιολόγηση τη Επιτροπή είναι επίγουσα η κατάσταση και ανησυχεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ασφάλεια και για τι ε, συνθήκε στην καμπανία. Γιατί ακολουθήθηκε η συνήθις διαδικασία και δεν ξεκίνησε μια εσπευσμένη διαδικασία, ούτως ώστε να ανακουφιστεί η περιοχή από την κατάσταση αυτή. Και άκουσα από τους αναφέροντες και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε σήμερα εδώ για να σας ακούσουμε, να μας τα λέτε εδώ ζωντανά. Γιατί πραγματικά είναι πολύ χρήσιμο το να βλέπουμε τους ίδιους τους ανθρώπους εδώ να μας τα λένε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Μιλήσατε για φιλμ και για ντοκιμαντέρ που δίνουν στοιχεία για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην καμπανία. Έχει γίνει όμως και έρευνα, επιστημονική έρευνα, που να δίνει αποδεικτικά στοιχεία. Έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρευνα για τους κινδύνους ε, για την ασφάλεια και για την υγεία στην καμπανία. Και κλείνω την παρέμβασή μου. Φαίνεται ότι υπάρχουν και νόμιμες και παράνομες ε, χωματερές και θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η διαφορά στην αντιμετώπιση των νόμιμων τόπων απόθεσης αποβλήτων και των παρανόμων. Πώς θα χειρίζεται η Ιταλική κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος κυρία Ντεμπρούν. Παρακαλώ να είστε πάρα πολύ σύντομοι, διαφορετικά δεν πρόκειται να τελειώσουμε. Yes, I'll use a shorthand version and hopefully the Commission will be able to understand. Θα είμαι πολύ σύντομη γιατί δεν έχουμε το χρόνο. Μόνο για, το, για την αναφορά 372 θα ήθελα να μιλήσω για την ατσέρα. Και ίσως να χρειαστεί να επανέλθουμε για το θέμα αυτό κάποια άλλη στιγμή. Αυτό το θέμα του 7% του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ε, που ε, λαμβάνεται από, την ανανεώσιμη, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και που χρησιμοποιούνται τα χρήματα για την καύση των ε, απορριμμάτων. Μας, ότι, μας είπαν ότι δεν υπάρχει ένδειξη χωριστά για το πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα χρήματα. Ποια είναι η θέση σας για αυτό το θέμα. Δεύτερον, όπως ακούσαμε από τους αναφέροντες, δεν έχει ανταποκριθεί η Ιταλία στις απαιτήσει της νομοθεσίας περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θα ήθελα να μας πείτε πώς έχει η κατάσταση ε, εφόσον ε, τροφοδοτούνται στον ε, αποτεφρωτή όλα τα απόβλητα. Δεν τηρούνται και τα δικαιώματά τους για πληροφόρηση και ενημέρωση. Ακούσαμε επίσης και για τα επίπεδα διοξινών, επίπεδα πολλών επιβλεβών ουσιών που τα υπερβαίνουν κατά πολύ τα στοιχεία που έχουμε από την Ιταλία. Ευχαριστώ, αλλά δεν έχουμε το χρόνο, γι' αυτό προσπάθησα να είμαι πολύ σύντομη. Αν θέλετε να σας τα ξαναπώ αναλυτικά αργότερα. Ε, παρακαλώ να είστε σύντομοι. Για όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν, ε, δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία ακούσαμε. Απλώς να τονίσω ότι πραγματικά είμαι έκπληκτη. Είναι πραγματικά σουρεαλιστική η κατάσταση που μας περιγράφεται μια κατάσταση σουρεαλιστική στην εποχή που ζούμε και εγώ που είμαι καινούρια ευρωβουλευτήνα και νέα στην ηλικία, εκπλήσωμαι που υπάρχει μια τέτοια κατάσταση σε μια χώρα όπως η Ιταλία. Πώς είναι δυνατόν. Με σοκάρουν αυτά που άκουσα. Και με σοκάρει το ότι υπάρχει ένα πολιτικό παιχνίδι πίσω από όλα αυτά. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι όλα αυτά μέσα στο παιχνίδι. Αλλά πώς είναι δυνατόν, πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση μέσα στα τελευταία δέκα χρόνια. Σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι το συντομότερο δυνατόν να, να, να ασχοληθούμε με αυτή την κατάσταση για να φροντίσουμε το αύριο αναφέρθηκαν θέματα δημόσιας υγείας που έχουν σχέση με τους χώρους διάθεσης αποβλήτων, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και τα μελλοντικά προβλήματα υγείας και δημόσια υγείας που θα έχουν σχέση με τη διαχείριση των, που, των αποτεφρωτήρων που δεν τηρούν τις προδιαγραφές και τις προδιαγραφές για τις εκπομπέ και ούτω καθεξής. Γιατί δεν λάβαμε μέτρα νωρίτερα. Χαίρομαι που ακούω ότι η Επιτροπή ε, θέλει να τηρούνται οι κοινωτικέ διατάξει. Εξάλλου, ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ακριβώ αυτό να είναι θεσμοφύλακα των συνθήκων. Δεν μπορεί να είναι αδύναμη η Επιτροπή να εφαρμόσει την κοινωτική νομοθεσία. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να υποχρεώσει μια χώρα παρότι υπάρχει διαδικασία επιβολής μέτρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αν δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποχρεώσει λοιπόν μια χώρα, μπορεί να χρησιμοποιήσει οικονομικά μέσα. Μέσω της διάθεσης κονδυλίων από τα διαφορετικά ταμεία, ενισχύσεων για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Από τη στιγμή που ένα κράτος μέλος δεν παίζει σωστά το παιχνίδι, ένα από τα μέσα που μπορεί να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η απειλή οικονομικών επιπτώσεων και απειλή της διακοπής κάθε κοινοτικής ενίσχυσης προς αυτό το κράτος ή προς αυτή την περιφέρεια. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να, είναι, να φαίνεται παράδοξο αυτό, γιατί μια χώρα που χρειάζεται πόρους για να λάβει αποφάσεις και να βελτιώσει την κατάστασή της, λέμε ότι ε, μπορούμε να τις στερήσουμε αυτά τα κονδύλια και μπορεί να ακούγεται παράδοξο. Παρ' όλα αυτά, ε, εδώ ε, είμαστε σε μια κατάσταση παραλόγου. Αν μετά από 10 χρόνια η Ιταλική κυβέρνηση δεν δείχνει να καταλαβαίνει, ε, ας ακολουθήσουμε πιο ακραία μέσα. και πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια, γι' αυτό να κρατήσουμε την αναφορά αυτή ανοιχτή και αν δεν μπορούν οι πολίτες ε, να λαμβάνουν πληροφόρηση από τη χώρα τους, θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τους εξασφαλίσει αυτή την ενημέρωση και η, Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει τις πληροφορίες αυτές από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ, κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, τις σύντομες παρατηρήσεις. Καταλαβαίνω τα αιτήματα των αναφερόντων. Στον 21ο αιώνα πρέπει να είμαστε σε θέση να επιλύουμε τέτοια προβλήματα. Natürlich müssen wir aufpassen. Wir haben auf Kein translation? No translation. The interpreters. Deutsch ist weg. Are going. Can you speak in English? In English. Perhaps. No. Ε, Δυστυχώ η διερμηνία διακόπτεται γιατί έχει ξεπεραστεί το όριο των 6,5. Geht's? Die gehen nach Hause, ja. Ja, sie, sie sind. I won't say when we have to go to Italia. We have to, to prepare this trip very, very uh, good. Uh, the petitioner, they won't help, and, and not only good words. As we have